Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ώρα νομίζω να αρχίσουμε. Άκουσα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ε, για εκείνους που ήρθαν με το αυτοκίνητο. Ε, ορισμένοι θα αργήσουν δηλαδή. Αλλά είναι αρκετοί συνάδελφοι εδώ. Έχω αποφασίσει να ξεκινήσουμε με την έκθεση της ΣΥΝΓΕΣ. Α, έχουμε όμως κάποια κατάλοιπα λίγο από χθε. Ο Ράιμερ Μπέργκερ. Μας έκανε εισαγωγή των θεμάτων που τον απασχολούσαν. Κανένας όμως δεν είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει, επειδή έλυγε η συνεδρίασή μας. Μου ελέγχθη τώρα ότι τουλάχιστον ε, μία συνάλληφο θέλει να αντιδράσει. Σας λέω όμως αμέσως ότι οπωσδήποτε στις 9.30 θα κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Άσχετα αν έχω ακόμα ολόκληρο κατάλογο ενδιαφερομένων ή όχι. Θα συνεχίσουμε αργότερα. Έτσι και αυτό είναι θέμα που θα συζητήσουμε πολύ συχνά. Λοιπόν, 10 λεπτά. Παρακαλώ. Sí, muchas gracias, Yuta. Ναι, ευχαριστώ πολύ Γιούτα. Θα κάνω μια απόπειρα να είμαι σύντομη και πολύ ακριβής στα σχόλια που θα κάνω για αυτά που συζητήσαμε χθες εδώ. Κρίμα που δεν είχαμε χρόνο να το συζητήσουμε χθες, διότι θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέγκε για την προσφορά που έκανε προς όλες τις ομάδες για να συνεργαστούμε, αλλά δεν κατάλαβα καλά τι ακριβώς πορεία σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε μετά από την προφορική ερώτηση και ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Εχθές ο κύριος Λαμασούρ έλεγε ότι ο στόχος τον οποίο πρέπει να επιτύχουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο συμμερίζομαι πλήρως είναι να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο, όχι με τους πρέσβεις, διότι εκεί μιλάμε για τεχνικές ε, διαπραγματεύσεις, αλλά μια πολιτική συμφωνία. Και εφόσον είναι σαφές ότι αυτή, αυτός είναι ο στόχος μας, να επιτύχουμε αυτή την πολιτική συμφωνία και αυτό που θέλουμε εμείς ως ε, ε Κοινοβούλιο, αλλά θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, είναι να βρούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτές τις νέες προτεραιότητες, για τις νέες ανάγκες που έχουμε θα πρέπει να τις ποσοτικοποιήσουμε. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγα τα πράγματα. Διότι άλλο είναι να προσπαθούμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση για ένα δίσε για παράδειγμα, ε, αυτά τα οποία προσπαθούμε να δώσουμε στο ε, μέσο ευελιξίας, ε, και άλλο να πούμε ότι θέλουμε δύο δις δεν χρειάζεται να είμαστε ακριβείς με το τελευταίο σέντ, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε λίγο την τάξη μεγέθους για να μπορέσουμε να ξέρουμε και τι άγουσα θα ακολουθήσουμε και ποια θα είναι η στρατηγική η οποία ε, πρέπει ε, να υιοθετηθεί. Και νομίζω ότι αυτό που κατάλαβα χθε από την παρέμβαση του κυρίου Μπέγκε είναι ότι η πρόθεσή του είναι να φτάσει μέχρι τέλους και με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα να μην εγκρίνουμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, ε, όχι τις επόμενες ακριβώς, αυτές που πρέπει να εγκρίνουμε και να μην τις ε, νομιμοποιήσουμε, διότι θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτού. Ε, δεν έχουμε μεγάλο περιφόρο ευελιξίας, αλλά μπορούμε να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε. Και αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Δεν ξέρω αν θα είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε μέχρι τέλους με αυτό, αλλά όπως και να έχει, ο στόχος θα πρέπει να είναι σαφής και όπως έλεγα και η στρατηγική μας. Ανεξάρτητα από τη θέση που θα μπορούσαν να έχουν αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να είναι αρκετά σαφής, θα πρέπει να καθορίσουμε εμείς τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν θα παρέμβει κάποιος άλλος ή κάποια άλλη πολιτική ομάδα, αλλά θα ήθελα να διαγράψουμε λίγο την πορεία μας διότι εχθές δεν κατάλαβα πολύ καλά τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, προς τα πού πάμε. Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Nein. Reimer, möchtest du daran... Ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Ράιμερ, θέλεις να απαντήσεις. Νομίζω ότι όσον αφορά τους βασικούς προσανατολισμούς, συμφωνούμε. Τώρα, το σε ποιο επίπεδο θα γίνουν οι συζητήσεις και οι αυτό δεν αφορά τον τριμερή διάλογο, γιατί ήταν πάντα η Προεδρία σε επίπεδο τουλάχιστον Υπουργού, τουλάχιστον, τουλάχιστον όμως ε, Υφυπουργού εκπροσωπότητα. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην ε, ε, διαδικασία συντονισμού που θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Εκεί ποιον θα έχουμε. Το είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρος μας ότι εκεί θα έχουμε μια άλλη δομή του εκπροσώπησης του Συμβουλίου για να μπορούμε να έχουμε μια πραγματική πολιτική διαπραγμάτευση. Εκτός αυτού θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα χθες και στη συζήτηση για την προφορική ερώτηση. όλα αυτά δεν ωφελήσουν τελικά. Υπάρχει και το άρθρο 324 του Συνθήκης του Λισαβόνας, όπου λέγεται ότι υπάρχει δυνατότητα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλεί τον πρόεδρο του Συμβουλίου, Συμβουλίου όχι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τακτικές διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε σε αυτό το επίπεδο να μπορέσουμε να πετύχουμε την επίλυση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ε, πολιτική προπολογισμών. Ίσως και σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Όχι λύσουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε μια συμπληρωματική ε, πολιτική διάσταση. Και να πούμε ότι και το Κοινοβούλιο έχει κάποιες προσδοκίες και το θέμα ακριβώς των ποσοστών είναι αυτό το θέμα των αριθμητικών στοιχείων. Ακούσαμε δεν μπορούμε να ορίσουμε αριθμού, αριθμητικά στοιχεία, ε, Πρώτου, πάρουμε απόφαση. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πάρουμε την απόφαση όταν δεν ξέρουμε τι θέλουμε, τι θα γίνει με τον Γαλιλαίο, <coughs> ποιο θα είναι ο προπολογισμό για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει το 2012-2013. Πάλι θα έχουμε ένα διορθωτικό προπολογισμό και μετά θα υπάρχουν αναθεώρησεις. Δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, κάποιους προσανατολισμούς και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν διάφορες ιδέες, θα πρέπει να παρουσιαστούν για να βρούμε και μια πολιτική λύση, ούτως ώστε να μην χρειάζεται τρία χρόνια, σειρά τρία χρόνια, να εξετάζουμε τι θα κάνουμε και που θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Γιατί αν δεν βρούμε τη λύση θα είμαστε επί τρία χρόνια στα μαχαίρια. Λοιπόν, το θέμα των της ποσοτικοποίησης, το θέμα των προτεραιοτήτων και μετά η πολιτική απόφαση του τι θα χρηματοδοτήσουμε τώρα και ποια είναι τα μέσα που έχουμε. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβάλλουμε και κάποια μέσα για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, εάν αυτό το 003 δεν επιληθεί επαρκώς, δεν θα χρειαζόμαστε να σκεφτόμαστε την αναθεώρηση τα επόμενα χρόνια, γιατί πάντα θα υπάρχει ένα κράτο που δεν θα συμφωνεί. Αυτό είναι ουσιαστικό για τι διαπραγματεύσει. Θα πρέπει εκ μια αρχή να ξέρουμε ότι δεν προτιθέμεθα να ε, υστερήσουμε εναντί αυτού που υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Πάντα να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε με την ισχύουσα διαδικασία να λειτουργήσουμε σωστά μέχρι αυτό το επίπεδο ούτω ώστε να μην μπορεί ένα κράτος μέλος να παρεμποδίσει την εξέλιξη. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε αυτές τις προϋποθέσεις και να πούμε τι θέλουμε να, να επιληθεί μέσω των διαπραγματεύσεων. Και αν μέχρι την Ολομέλεια δεν έχουμε συμφωνήσει η ψηφοφορία που θα γίνει το Σεπτέμβριο, αν δεν υπάρχει καμία κίνηση σχετικά με τις προτάσεις από την Κομισιόν, ή την προσφορά του Συμβουλίου, τότε πράγματι προτίθεμαι, εάν με υποστηρίξει πάνω σε αυτό η Επιτροπή, μας εδώ να πάω στην Ενωμένα και να πω απορρίπτουμε όλες τις προτάσεις. Και παρακαλούμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο να μας υποβάλουν νέες προτάσεις. Δεν μπορούμε έτσι να λειτουργήσουμε. Αλλά μόνο εάν το αποφασίσουν αυτό οι πολιτικές ομάδες. Για να παραμείνει η δέσμη όσα έχει και να μην επιτρέψουν στο Συμβούλιο ή στην Κομισιόν να μας φάνε μπουκιά-μπουκιά όπως υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση. Μπορούμε να σημειώσουμε αυτό που είπε ο Ράμερ Μπέγκερ, να αφήσουμε τη δέσμη ως έχει, δεμένη, να μην είναι οι πολιτικές ομάδες, όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι ενωμένο και αυτό που μας περιέγραψε και που είπε θα πρέπει να έχουμε λογικές καλές διαπραγματεύσεις ξέρουμε ότι δεν, χρειάζ, δεν χρειάζεται να κάνουμε έκκληση στην λογική του Συμβουλίου θα πρέπει να δείξουμε εμείς μια σταθερή στάση και ισχυρή στάση ούτως ώστε να μην μειώσουν τα δικαιώματα και τι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε ούτε πεντάρα για την λογική του Συμβουλίου. Ίσως αν είχαμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σαν ε, διαπραγματευτές, ίσως κάτι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά αν έχουμε τώρα τη διοίκηση του Συμβουλίου. Καθήκαμε. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Και ακριβώς για ένα σημείο προσπαθούμε να κινήσουμε το Συμβούλιο να μην υστερήσει σχετικά με το, τα διδασμένα του Κοινοβουλίου μέχρι στιγμής. το λόγο. Για να δω για το 8 μου λέτε να μιλήσω τώρα. Ωραία. Δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζει το Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Κομισιόν υπέβαλε πολύ φιλόδοξη πρόταση όπου πρόκειται να διατυπωθούν τα μισά άρθρα περίπου. Το αποκαλεί στα αγγλικά recast η Κομισιόν. Έχουμε πραγματικά τώρα πια όλα τα στοιχεία στα χέρια μας για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και χαίρομαι γι' αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν. Ελπίζω μέχρι τα τέλη του έτους να μπορέσει να υπάρξει η έκθεση. Είναι τεράστιο το έργο. Όλοι καλούνται να συνεργαστούν γι' αυτό, αν θέλουν. Γιατί θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα κείμενο και να προσπαθήσουμε έτσι να πραγματοποιήσουμε το όνειρο του να έχουμε ένα προπολογισμό μονολυθικό αν θέλετε. Το θέμα ότι πρόκειται για μία νέα μορφή του κανονισμού αυτού μας ε, προβληματίζει λίγο γιατί υπάρχει ένας ενδοθεσμικός ε, κανονισμός, μια συμφωνία μάλλον από το 2001, σύμφωνα με οποίο το Κοινοβούλιο ανέλαβε την υποχρέωση στην περίπτωση αναδιατύπωσης να ασχοληθεί μόνο με τα άρθρα με τα οποία έχει ασχοληθεί η Κομισιόν. Τώρα όμως οι στόχοι απλούστευσης ίσως καθιστούν ε, υποχρεωτικό να εξετάσουμε και άλλα σημεία Δηλαδή η νέα μορφή αυτή, εάν δεν άπτεται όλων των άρθρων, τότε δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι έχουμε εμεί κατά νου και τι έχει η Κομισιόν. Γιατί αν είμαστε δεσμευμένοι να εξτάσουμε μόνο τα άρθρα τα οποία έχει τροποποιήσει η ίδια η Κομισιόν, θα πρέπει να καθυστερήσουμε την πρώτη πρόταση για τη Λισαβόνα μέχρι το τέλος, ούτω ώστε μετά να εξετάσουμε εκείνα τα άρθρα τα οποία μου φαίνεται ότι θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Συνεργάζομαι με τον κύριο Ρεβελίνη, τον ε, εισηγητή στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Προσπαθούμε να καλέσουμε όλους να συνεργαστούν. Ε, σε αυτό το νέο θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των ε, εθνικών δηλώσεων, το θέμα του ανοιχτού κινδύνου. Προσπαθούμε με την Κομισιόν να τα εντάξουμε και τα στοιχεία αυτά στην δική μας πρόταση. Έχουμε λοιπόν κατά νου κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο, αλλά έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να έχουμε μία μονολογική, όπως σας είπα, πρόταση επιτέλους. Είχαμε ήδη μία ακρόαση πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, γραμματεία, να ευχαριστήσω και Σοσιαλιστική και την, την ομάδα των φιλελευθέρων, γιατί είχαν πάρα πολλούς ε, ομιλητές ορίσει και μπορέσαμε έτσι να ακούσουμε απόψεις της ε, κοινωνίας των πολιτών. Εγώ είχα αναθέσει και κάποιες μελέτες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μεγαλύτερη απλούστευση. Το πρόβλημα είναι ότι το θέμα είναι πολύ πολύ πλοκό και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε τα διάφορα ε, στοιχεία που υπάρχουν εκεί να τα συνενώσουμε. Είμαι πάντως αισιόδοξη ότι θα έχουμε μια καλή πρόταση τελικά. Θα μπορέσουμε να εισαγάγουμε τις απλουστεύσεις που έχουμε κατά νου. Δεύτερη μας ερώτηση προς την Κομισιόν είναι η ο κανόνας μας απλούστευσης με λιγότερους κανόνες μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Κατά πόσον δηλαδή μπορούμε να ορίζουμε τα πολιετή προγράμματα μετά το 2004. Αυτό θα ήταν 14, συγγνώμη, αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο καθένας όμως γράφει τα δικά του στοιχεία, τότε δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτά είναι που με απασχολούν. Τι κάνει η Κομισιόν εσωτερικά για να εξασφαλίσει ε, ο δημοσιονομικός κανονισμός να τηρεί όλους αυτούς τους κανόνες που προανέφερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν που έχει στήσει το λόγο εδώ και γι' αυτό μπορούμε αμέσως να περάσουμε σε εσά, κύριε Γενική Διευθυντά. Ακούσατε φαντάζομαι τις ερωτήσεις της κυρίας Γκρέσλε. Καταρχήν πρέπει η Κομισιόν να μας ορίσει τι σημαίνει το recast που λέει. Και δεύτερον θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την απλούστευση των κανόνων και κατά πόσον δεν θα έχουμε επικαλύψεις. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις της κυρίας Γκρέσλε. Έχω μπροστά μου το έγγραφο στη γαλλική γλώσσα, το οποίο λέγεται «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το δημοσιονομικό κανονισμό για τον προϋπολογισμό των γενικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Είναι σαφές ότι οι προτάσεις αυτές αφορούν κάποια συγκεκριμένα άρθρα του ισχύοντος κανονισμού έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν αυτό το οποίο ονομάζουμε στα αγγλικά accountability, δηλαδή το να είναι κάποιος υπόλογος και την υπευθυνοποίηση θα έλεγα στα πλαίσια του συνδυασμού των πόρων και της σωστής τους χρήσης. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σαφές ή θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σαφές για μας, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρήσει ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποιήσεις σε άλλα τμήματα. Θα τα επανεξετάσει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο τέλος της διαδικασίας θα δει αν χρειάζεται να τροποποιήσει τη διαδικασία αυτή. Θα τεστεί λοιπόν το θέμα αν η Επιτροπή σας είναι διατεθειμένη να κάνει και αυτή κάποιες αλλαγές στις προτάσεις της στα πλαίσια βέβαια του σεβασμού των σταδίων της διαδικασίας που είναι αρκετά περίπλοκη στην περίπτωση της συναπόφασης. Δεύτερον, σχετικά με το όνειρο ε, για απλούστευση, την απλοποίηση της κυρίας Γκρέσλε, προφανώς και το σημεριζόμεθα Και ο παρακαθήμενος συνάδελφος και εγώ Έχουμε βάλει αυτόν τον στόχο της απλοποίησης. Θέλουμε να καταστήσουμε τον κανονισμό αυτό ε, φιλικό προς τους χρήστες, user-friendly. Θέλουμε να τον καταστήσουμε εύκολο στην χρήση από τους εισαγωγικά πελάτες, τους χρήστες. Αυτό είναι ακριβώς που βρίσκεται στο κέντρο, θα έλεγα, των ανησυχιών μας. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα προόδου, φυσικά πάρα πολλά μένει να γίνουν αλλά νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος. Τίθεται τώρα το θέμα της σχέσης ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχουμε ήδη κάνει γύρω από τον κανονισμό αυτό και τους λεγόμενους τομεακούς κανονισμούς, τους το κανονισμούς κατά τομέα. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Βασικός μας στόχος του Επιτρόπου Λεβαντόφσκι δηλαδή και της Γενικής Διεύθυνσής μας είναι να υπάρξει μία κάποια συνοχή ανάμεσα σε αυτά τα οποία θα προχωρήσουμε να κάνουμε στα πλαίσια του Γενικού Δημοσιονομικού Κανονισμού και από την άλλη στους τομεακούς κανονισμούς. Γιατί αν δεν το πετύχουμε αυτό αμφισβητείται η χρησιμότητα της παρέμβασής μας. Δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω τίποτα το ιδιαίτερα εμπιστευτικό, αλλά ο στόχος αυτός είναι κάτι το οποίο έχει, θα έλεγα, εντοπιστεί από τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι στα πλαίσια της υιοθέτηση των προτάσεων από το σύνολο των Επιτρόπων της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω τη λέξη να διαβεβαιώσω την κυρία Γκρέσλε να αντισπούμε πούμε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα και ο ίδιος ο Επίτροπος και το σύνολο των Επιτρόπων κινητοποιούνται γύρω από την υπόθεση αυτή και ε, η Γενική μου Διεύθυνση θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τη συνοχή ανάμεσα στους ε, κατατομείς κανονισμούς και τον γενικό κανονισμό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Τώρα έχουν δύο ακόμα ζητήσει στο λόγο, ο Γιάννη Κάιε και μετά ο Γιώργο Μιλφέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα ότι έχουμε δύο προτάσεις της Κομισιόν για την αλλαγή του δημοσίου κανονισμού δηλαδή την ε, τριετή αναθεώρηση των ε, θέματα της Λισαβόνας και αυτά που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εγώ αναρωτιέμαι κατά πόσον, κατά χρειάζεται να υπάρχουν τρεις διαφορετικές προτάσεις, ε, γιατί αυτό μας βάζει στο πρόβλημα να αναγκαστούμε να λύσουμε την ίδια παράγραφο περισσότερες της μιας φοράς να εξετάσουμε επίσης τις τρεις δέσμες και γι' αυτό αναρωτιέμαι κατά πόσον η Κομισιόν βλέπει να υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, ποια θα ήταν η στάση δηλαδή, εάν εν ώψη αναγκαιότητας της ε, γρήγορης ε, δημιουργίας της Επιτροπής Εξωτερικής, της Υπηρεσίας Γνώμη Εξωτερικής Δράσης, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ίσως από εκεί. Jürgen Το ίδιο θέμα θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ. Δεν ήμουν παρόν όταν συζητήθηκε το θέμα στα πλαίσια των συντονιστών. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί από τη μία μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλεονέκτημα συγκεντρώνοντας τα τρία τμήματα του πακέτου μαζί. Από την άλλη όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες σε σχέση με την εξωτερική υπηρεσία και ίσως αυτό το τμήμα του δημοσιονομικού κανονισμού καλό θα ήταν να το εντάξουμε στο πακέτο το σχετικό με την εξωτερική υπηρεσία. Και το ίδιο ισχύει επίσης και γύρω από τα θέματα της Λισαβόνας. Θα μπορούσε να είναι επίσης ένα τμήμα του πακέτου της Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καθυστερήσουμε άλλα σημαντικά τμήματα των πολιτικών μας για να κρατήσουμε συνεκτικά τα τρία τμήματα του ε, γενικού κανονισμού. Έλγα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στη γενική συζήτηση για το δημοσιονομικό κανονισμό είχα αναφέρει στην προηγούμενη μας συζήτηση. Τι γίνεται όσον αφορά την απλούστευση κάποιων κανόνων. Όχι να καλέσουμε κάποιον να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά ασυνείδητα ή να οδηγήσει σε ε, απάτες, τεσταλίες κλπ. Αλλά να προσπαθήσουμε να έχουμε ακριβώ κάποια διευκόνηση για τις μικρές ιδίως... Ε, προτάσεις για τα μικρά σχέδια, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί με καλές ιδέες που τους αποδιώκουμε γιατί ακριβώς ε, τους τρομάζει το πολύπλοκο των διαδικασιών. Και θα ήθελα σήμερα και από αυτόν να ζητήσω την Κομισιόν και την κυρία Γκρέσλε να μου πούνε την άποψή τους. Όσο σημαντική και αν είναι η γενική συζήτηση, αυτό το θέμα της απλούστευσης του δημοσιονομικού κανονισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας όσον αφορά την αποδοχή του από τους πολίτες. Ευχαριστώ. So, jetzt habe ich keine weiteren Wortmeldungen. Πρόεδρος, δεν έχει ζητήσει ακόμα κανένα άλλο το λόγο. Ίσως θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε στην Κομισιόν να απαντήσει στις ερωτήσεις που επιβλήθησαν. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω και την ε, αρχική ερώτηση της Κομισιόν, γιατί όταν απάντησε η Κομισιόν, εγώ δεν κατάλαβα να υπήρχε μια σαφής απάντηση. Γιατί δεν ετέθη το θέμα ότι θα πρέπει εκ των προτέρων να αναλάβει την υποχρέωση της Κομισιόν να δεχθεί τις τροπολογίες που θα υποβάλουμε εμείς. Το θέμα ήταν ε, η νομική αξιολόγηση και θα ε, ε, ήμουν πραγματικά ευχαριστημένη εάν ο Γενικός Διευθυντής άκουγε εμένα, όχι του συνεργάτες του. Λοιπόν, πρόκειται για το θέμα κατά πόσον εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε σε θέση άρθρα τα οποία η Κομισιόν δεν έχει τροποποιήσει μέσα στα πλαίσια αυτής της αναδιατύπωσης. Έχουμε λέω εμείς το δικαίωμα να τα εξετάσουμε και να τα τροποποιήσουμε ή μετά θα έρθει η νομική υπηρεσία της Κομισιόν και θα μας πει όχι, όχι, αυτό δεν προβλέπεται και γι' αυτό απογορεύεται. Αυτή ήταν η ερώτησή μας αρχικά. Θα ήθελα πάνω σε αυτό μια σαφή απάντηση και όσον αφορά επίσης ε, αυτό το θέμα των τριών τμήματων της τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα ήθελα απάντηση. Ναι, Πρόεδρε, σχετικά με το πρώτο σημείο. Δεν μπορώ να αναλάβω καμία δέσμευση σε αυτή τη φάση. Είπα όμως, ίσως λίγο συμβιλικά, αλλά νομίζω ότι το θέμα θα εξαρτηθεί από την ίδια την εξέλιξη της διαδικασίας της συναπόφασης. Όλα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το θέμα και κατά πόσον θα κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεπέμβει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν πράγματι δεν υπάρξει επιστροφή ή feedback <clears throat> προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν η διαδικασία είναι διαφορετική, τότε ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να εξετάσει τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. γύρω από τις τρεις διαφορετικές προτάσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Φέμ έχει δώσει μια σωστή περίληψη της υπόθεσης. Έχουμε διαφορετικού τύπου προσθεσμίες εδώ θα έλεγα. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα ε, ε επίγοντος για τον καθένα, για το κάθε όργανο. Το βασικό όμως είναι να έχουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις του κανονισμού στη διάθεσή μας, έτσι ώστε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να τεθεί σε λειτουργία. Αν δεν υπάρξει τροποποίηση, δεν θα υπάρξει υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Γιατί δεν υπάρχουν ε, προβλέψεις ε, για τον προϋπολογισμό, έτσι ώστε να λειτουργήσει η υπηρεσία αυτή. Είναι απλό. Επιμένουμε λοιπόν έτσι ώστε οι τροποποίησει στο δημοσιονομικό κανονισμό που είναι απαραίτητες για τη θέση σε λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης να γίνουν δεκτές πάρα πολύ σύντομα έτσι ώστε να εξετάσουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού της εξωτερικής υπηρεσίας και στην υιοθέτηση του προϋπολογισμού της εξωτερικής υπηρεσίας και να μπορέσει να λειτουργήσει η υπηρεσία αυτή από το φθινόπωρο και μετά. Τώρα 1η Οκτωβρίου θα γίνει αυτό, 1η Νοεμβρίου δεν ξέρω, κανείς δεν το ξέρει πάντως. Αυτό που ξέρω είναι ότι όλες αυτές οι προβλέψεις είναι απαραίτητες για να τεθεί σε λειτουργία σε εύθετο χρόνο η υπηρεσία εξωτερικής δράσης σχετικά με την τεχνική προσαρμογή στη συνθήκη, πάνω κάτω ακολουθούμε την ίδια προβληματική. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη να επιτρέψουμε σε όλους τους εμπλεκομένους να καταστούν ικανοί και να μπορέσουν να ωφεληθούν από τις πρόοδους οι οποίες έχουν επιτελεστεί στα πλαίσια της νέας συνθήκης. Εάν δεν υπάρξει μια τροποποίηση των προβλέψεων του δημοσιονομικού κανονισμού για να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της Λισαβόνας, δεν θα τεθούν σε λειτουργία οι παρατηρήσεις αυτές. Και νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνει τα απαραίτητα έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να τεθούν σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν, γιατί αλλιώς παραμένουμε στις παλαιές προβλέψεις της συνθήκης και της διοργανικής συμφωνίας κάτι το οποίο θα δημιουργήσει θέματα στη καθημερινή διαχείριση του προϋπολογισμού. Γνωρίζουμε όλοι επίσης ότι οι συζητήσεις οι σχετικές με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σχετικές επίσης με κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην μεγάλη σε εισαγωγικά πρόταση τροποποιήσεων που έχουμε κάνει, οι συζητήσεις αυτές απαιτούν χρόνο και είναι πιθανό να πρέπει να περιμένει κανείς περίπου δύο χρόνια. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε εμείς τόσο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο χρόνο για τη θέση σε ισχύ ε, ε, και σε λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και δεν νομίζω ότι είναι καν προς το συμφέρον των θεσμικών οργάνων να περιμένουν δύο χρόνια έτσι ώστε να τεθούν σε λειτουργία οι τεχνικές ρυθμίσεις που απορρέουν θα έλεγα από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίληψη που έχουμε. Ίσως η αντίληψη αυτή να μην, είναι, να μην μεταφέρει ένα τεράστιο ενθουσιασμό, αλλά είναι θα έλεγα μια αντιμετώπιση των πραγμάτων πρακτική, αποτελεσματική και επιτρέπει στα όργανα να δουλέψουν, να δουλέψουν γρήγορα, να δουλέψουν αποτελεσματικά. Ja, vielen Dank. Ähm. Ευχαριστώ. Μου υπενθυμίζουν και θέλω να υπενθυμίσω και ο συνάδελφους ότι στις δηλώσει μας θέλουμε να, λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τα πάντα ούτως ώστε το των δυνατόν όλα όσα σχετίζουν με τη συνθήκη της Λισαβόνας να εφαρμοστούν. Και μεταξύ αυτών είναι βέβαια και το ότι θα πρέπει η υπηρεσία εξωτερική δράση και όλε οι άλλε επιπτώσει από τη συνθήκη τη Λισαβόνα να μπορέσουν το γλυγορότερο δυνατόν να εφαρμοστούν. Η Ίγκεμποκ έχει το λόγο τώρα και μετά θα κλείσουμε αυτό το Σελβατόρ. Um, Και μετά θα κλείσουμε λέω το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που άκουσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να ε, πάρω όμοιρο αν θέλετε την πρώτη ε, αναθεώρηση της Λισαβόνας για να μπορέσουν να περάσουν τα άλλα σημεία γιατί αν δεν υπάρχει καμία δέσμευση της ε, Κομισιόν θα είμαστε ανεξάρτητοι για την τριετή αναθεώρηση δεν θα ήταν πολύ ευφυές ε, να δράσουμε διαφορετικά. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να καθυστερήσω. Του Ναντίνα. θα χαιρόμουν να τελειώσουν τα πράγματα, αλλά εδώ θα πρέπει να προσπίσω τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε η Κομισιόν της διαδικασίε, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε σήμερα αυτά που είναι για μας σημαντικά. Η πρώτη αναθεώρηση λοιπόν θα αφορά οπωσδήποτε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από το να εξετάσουμε το σύνολο της δομής. Δεν μπορώ να επιβάλλω έναν έλεγχο εάν δεν ξέρω ποια είναι η δομή. Φαντάζομαι θα μπορέσουμε εδώ να συνεχίσουμε. Και η ερώτηση που υπευλήθη αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικά. Το άρθρο 1, παραδείγματο χάρη που αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα τροποποιηθεί τρει φορέ. Εγώ ήθελα να το αλλάξουμε μία φορά το άρθρο αυτό, στην τωρινή αναθεώρηση, και να εγγράψουμε αυτό που αρμόζει να εγγραφεί. Δηλαδή, ότι πρέπει να πραγματοποιήσουμε όλα αυτά που αναφέρεται στην συνθήκη της Λισαβόνας, για να μην χρειαστεί να επανέλθουμε στην τριετή αναθεώρηση. Δηλαδή, θα λέει ότι όλα τα θεσμικά όργανα που αναφέρονται στην συνθήκη της Αβώνας και η υπηρεσία εξωτερικών δική δράσης θα αναφέρονται στο άρθρο 1 για να μην επανερχόμαστε συνεχώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να έχουμε, σύμφωνα με τις δυνατές μας, διευκρίνηση του τι κάνουμε εδώ. Για τη Λισαβόνα την ίδια διαδικασία είναι σαφής. Αυτά που έχουμε συμφωνήσει δεσμεύουν όλους. Δεν τίθεται θέμα. Τώρα από νομικής απόψης πώς μπορώ να πετύχω απλουστεύσεις είναι ένα θέμα σημαντικό και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η πρόταση Λισαβόνα. Και γι' αυτό λέω ότι θα πάρουμε όμοιρο αυτή τη συνθήκη γιατί δεν μας δίνει άλλες δυνατότητες η Κομισιόν. Εάν μας προτείνει κάτι διαφορετικό θα μπορούμε να δράσουμε και εμείς διαφορετικά. Κυρία Τρίπελ, την τελευταία αναθεώρηση προβλέψαμε ήδη μία κοινοποίηση στους δικαιούχους. Πολλά απλουστεύτηκαν έτσι, αλλά βέβαια δεν αρκούν ακόμα. Έχουμε πάλι το πρόβλημα ότι οι μικροί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις πολλές προτάσεις. Και είδαμε ότι εκεί που δεν έχουμε εμείς διατάξεις, θεωρεί η Κομισιόν ότι είναι δική της η πρόταση. Δηλαδή εκεί όπου εμείς προβλέπουμε μία απλούστευση εθελοντικά δεν προωθείται. Κάναμε πολλά για απλούστευση. Αν δω όμως τον τομέα της έρευνας, τα προβλήματα που έχουν, ε, τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε είναι οι τόκοι για την προχρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Και αυτή τη στιγμή εξαρτώμεθα η Κομισιόν να το επιβάλλει ίδια. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στο προπολογισμό είναι στα ειδικά ταμεία, με διάφορα που υπάρχουν εκεί και αν δεν μπορεί εσωτερικά να το διευκρινίσει η Κομισιόν, τότε δεν θα μπορέσουμε κι εμείς μόνοι μας να πετύχουμε τίποτα. Γι' αυτό θα ήταν σημαντικό κύριε Γενική Διευθυντά να προχωρήσουμε εδώ. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να είμαστε καλύτεροι στο μέλλον από ό,τι είμαστε ήδη. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ καταρχήν τη συζήτηση του σημείου αυτού και περνάμε τώρα στο σημείο 19. που πρόκειται για ενημέρωση της ε, υπηρεσίας για ανταγωνιστικότητα και καινοτομίες, η οποία θέλει να τη δώσουμε το πράσινο φως για να το πω έτσι, να υπογράψει ένα, μια σύμβαση για ένα κτίριο. Η Μόνικα Χολμάιερ είναι συγγετριά. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, για το θέμα αυτό του κτηρίου για το ΕΑΣΕΗ προσπάθησα να δώσω τα, όλα τα κείμενα στον συνεισηγητή. Ήταν ογκώδες ο φάκελος, αλλά βλέπω όμως ότι πολλές φορές χρειάζεται να επιμείνουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να μάθουμε το συγκεκριμένο κόστος για το προϋπολογισμό. Λίγα λίγα μας το δίνουμε το σταγονόμετρο. Λοιπόν, πρώτη για την υπηρεσία αυτή η οποία δημιουργήθηκε το 2003 και από το 2006 και μετά είχε κάποια γραφ... γραφεία σε ένα κτίριο στο λεγόμενο κτίριο Madu Towers, 66.000 ευρώ το χρόνο. Μετά υπήρχε ένα άλλο κτίριο που νίκιασαν στο Square Fair Orba. το οποίο κόστησε 415 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο ήταν ε, σχεδόν 800.000, 415.000 συγγνώμη, το σύνολο των 800.000. Ε, πρόκειται για μια μεταβατική λύση γιατί ε, το κτίριο στην Σκουέφρα Ρόμπαν πρόκειται έτσι και να κατεδαφιστεί όταν ε, αποσυρθεί από εκεί η υπηρεσία μας. Υπήρξαν τρεις διαγωνισμοί συνολικά. στο τελευταίο διαγωνισμό υπήρχαν 26 προσφορές, οι δύο από αυτές ήταν σύμφωνες με όλα τα κριτήρια και βάσει αυτών επελέχθη το σχέδιο του κτίριου που έχουμε αυτή τη στιγμή που είναι για την Place Rogier 16 ο ιδιοκτήτης είναι η μομπλία του Royal Rogier SS πρόκειται για την εκμίσθωση 6.499 τετραγωνικών και 15 θέσεις ε, σχόλους και υπάρχει μία σύμβαση ετήσιας μίσθωσης 1.116.340 ευρώ και κόστος για, την, ε, για τον εξοπλισμό Υπάρχει το λεγόμενο κόστος του εξοπλισμού fitting out που συμπεριλαμβάνει και κτίρια και πόρτες και τέτοια. Γιατί τώρα πια νοικιάζουμε κτίρια στα οποία πραγματικά τα χτίζουμε σχεδόν. Έτσι λοιπόν το τελικό κόστος είναι κάπως υψηλότερο. Το κτίριο αυτό κατά τη μου βρίσκεται σε πολύ καλή θέση. Είναι εκτός ε, του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής γειτονιάς, ε, περίπου 3 χιλιόμετρα από τον Περλεμό, καλά συνδεδεμένα. Υπάρχουν τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας. Και μπορούσα επίσης να δούμε ότι υπάρχει ήδη μια καφετήρια γιατί ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα, ένα, μια άλλη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης ε, ε πληροφορική και ούτω καθεξής. Ε, η, συνδίκη προβλέπει, η σύμβαση προβλέπει 15 χρόνια. Βέβαια θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει η υπηρεσία αυτή ε, τα επόμενα 15 χρόνια. Θα πρέπει να το κατά πάσα πιθανότητα θα τη χρειαστούμε. Έτσι το κόστος νομίζω ότι είναι εντάξει. Μετά, ε, πρέπει να εξάσουμε το θέμα του αμοιάντου. Έγινε κάποια έρευνα και υπήρχε κάπου αμοιάντος. Ανταλλάχθηκε αυτό το υλικό. Δεν υπάρχει λοιπόν πια αμοιάντος στο κτίριο. Ο προπολογισμό το 2010 και το σχέδιο προεπιλογισμού 2011 λαμβάνουν ήδη υπόψη το προσωπικό και την αύξηση της επιφάνειας γραφείων. Ξαναρώτησα, Πρόεδρε, γιατί η μέρη στις υπηρεσίες αυτές χρειάζεται να νοικιαστούν κτίρια που δεν λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη του αριθμού του προσωπικού. Και έτσι οι υπηρεσίες αυτές ε, αντιμετώπισαν κάποια στιγμή δυσκολίες. Θα πρέπει στο μέλλον ίσως να δράσουμε πιο προληπτικά. Μπορώ λοιπόν τώρα να θεωρήσω όμως ότι δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Ένα πρόβλημα υπάρχει αυτό το τύπο σύμβασης που αυξάνει το κόστος ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τη συντήρηση. Δηλαδή θα πληρώνουμε όχι μόνο τον νίκη αυτό καθευτό αλλά και την συντήρηση του κτηρίου. Αυτό το, την πληροφορία την πήραμε έτσι την τελευταία στιγμή. 1.495.000 είναι το κόστος αυτό. Αλλά βέβαια το θέμα της, ε, του εξοπλισμού και της μετατροπής ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε τις επόμενες μήνες γιατί αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται και μέσω διαγωνισμού, αλλά αναθέτηται σε κάποιον. Πρέπει να το κοιτάσουμε, γιατί στο κάτω-κάτω πρόκειται για 2,5 εκατομμύρια. Τούτο λεχθένος είμαι υπέρ του σχεδίου και όταν μου δώσουν τις ιδέες τους οι συνεισηγητές, μπορούσαμε νομίζω να προχωρήσουμε. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ Μόνικα. Νομίζω ότι πραγματικά εδώ θα πρέπει να εργαστούμε λιγάκι περισσότερο γιατί πάντα πιάσαμε την διοίκηση του Κοινοβουλίου να υπάρχει πάντα το σχέδιο διαχείρισης ε, προσωπικού κτίριου όλα μαζί και θα ήταν καλό και για την Κομισιό νομίζω να ε, υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Καρ Χάλπλουμ έχει δει το λόγο. Thank you, Mrs. Chair. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Έκανε για μια ακόμη φορά εξαιρετική δουλειά για να υπολογίσει το πραγματικό κόστος σχετικά με το κτηριακό. Η ιδέα γενικά φαίνεται καλή. και θα δώσει στην υπηρεσία το σωστό χώρο. Πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι όταν το τα κόστη για την ανακαίνιση τα φορτώνεται η ίδια η υπηρεσία είναι για 15 χρόνια το κόστος αυτό θα πρέπει να κατανεμηθεί δηλαδή ώσπου να αποσβεστεί ενώ η υπηρεσία αυτή προβλέπεται σε μια πρώτη φάση να λειτουργήσει μέχρι το 2015. Δεν έχουμε εγγυήσει για την ε, συνέχιση λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας. Λοιπόν, μακάρι να συνεχίσει, αλλά δεν υπάρχουν νομικές εγγυήσει. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει και προηγούμενο σχετικά με οικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες να παρατείνονται και μετά το τέλος της λειτουργίας μιας τέτοιας υπηρεσίας ή ενός τέτοιου οργανισμού. Πέραν αυτής της παρατηρήσεως όμως γενικά νομίζω ότι η απόφαση είναι σωστή. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, και αυτό θα πρέπει να γραφτεί ακριβώς στις κατευθυντήριες γραμμές. Γιατί ε, αυτές οι εκτελεστικές υπηρεσίες έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια. μπορεί κανείς να να βγει από το ε, συμβόλαιο μετά από πέντε χρόνια, με το καταγγείλει. Αυξάνεται όμω το νίκη βέβαια, γιατί υπάρχουν διάφορα κόστη που δεν αποσφύνονται πια σε 15, αλλά σε πέντε χρόνια. Αν πούμε εκ μέσα αρχής πέντε χρόνια δεν θα μα αφαιρώσουν ε, το κτίριο. Φαύλο κύκλο λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα δημοσιομικών κανόνων γενικά, γιατί ε, είδαμε ποια είναι τα κτίρια τα οποία ζήτησαν να εγκριθούν οι Κομισιόν και ποια όχι. Εκείνα που δεν έχουν εγκριθεί ε, είναι εν μέρει τεράστια και που δεν είχαν υποβληθεί ε, στην Επιτροπή Προπολογισμού. αυτό το σύστημα δηλαδή της υποβολής ή μη υποβολής εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εδώ το θέμα είναι ότι πρόκειται για μια εκτελεστική υπηρεσία και όχι μια υπηρεσία της Κομισιόν. Το είχαμε γράψει τότε στις διατάξεις για τις εκτελεστικές υπηρεσίες ότι οπωσδήποτε θα είναι υπό το δικό μας έλεγχο. Κτίρια, οτιδήποτε. Εν αντιθέσει από το πρέπει να κάνει κατά τα άλλη κομισιόν. Είμαι υπέρ των κατευθυντηρίων γραμμών. Δεν μπορεί να έχει κανένα ένα κανόνα για όλου, αλλά θα πρέπει να έχουμε τέλο πάντων κάποια περιθώρια ρημούλα όλους και οπωσδήποτε θα συστήριξουμε σε αυτό που είπες. θα πρέπει τώρα όμως να αποφανθούμε κατά πόσον θα ακολουθήσουμε την πρόταση της ηγήτριας και δεν θα γνωμοδοτήσουμε αλλά θα λάβουμε υπόψη αυτό που θέλει η υπηρεσία αυτή απλώς. Ποιος είναι κατά της πρότασης. Κανένας. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα προετοιμάσουμε εμείς καμία έκθεση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και αυτό το σημείο και περνάμε στις μεταφορές και στην ψηφοφορία. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω σε όλους τους συναδέλφους ότι ο Ρομπέρτο Καλτιέρη θα ξανάρθει εδώ στις 11 παρατέταρτο για να μας παρουσιάσει το χτεσινό αποτέλεσμα. Τώρα θα έχουμε την όλη της ψηφοφορίας και μετά θα ξα... ε, ε, ασχοληθούμε με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Haben wir Transfer. Ja, genau. Transfer νούμερο 16. Μεταφορά υπαριθμών 16, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. στο Kobe News ε, σημειώνονται πέντε μεταφορές. Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή για να πάρουμε αποφάσεις γύρω από το 16 και το 17 και να αφήσουμε τα άλλα τρία για απόφαση στην επόμενη συνάντησή μας. Η πρόταση αυτή μόλις έφτασε τώρα, πριν λίγες μέρες δηλαδή, μας έφτασε δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε κτλ. Και δεν μπόρεσα να έχω μέσα σε δύο-τρεις μέρες επαφές και με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Αλλά για το 16 και ίσως και από κοινού το 17 για να μην καθυστερούμε, εγώ σας προτείνω να δεχθείτε τις μεταφορές αυτές και τις δύο. Ίσως κάποιοι συνάδελφοι να έχουν απορίες, αλλά γενικά θα έλεγα ότι οι απαντήσεις θα γίνουν αποδεκτές και μπορούμε να τις υπερψηφίσουμε, τις 16 και 17. Υπάρχουν ερωτήσεις. Α, είναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ, πρόεδρε. Ήταν δύσκολο να έχει κανένας ε, πληρικό. Να το πρώτο κείμενο έχει 167 Σελίδε και δεν ήταν πολύ διαφανή η κατάσταση. Όταν προσπαθεί κανένα όμω κάτι καταφέρνει. Έχουμε τώρα και στοιχεία για Excel. Το 2005 και 2006 είχε δαπανίσει για τη κομισιών 608 εκατομμύρια ευρώ σε τέσσερα χρόνια. Εγώ δεν διαφωνώ με τη μεταφορά σήμερα, αλλά θέλω να μου απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις. Αν δει κανένα τα έγγραφα αυτά, τα βλέπει ότι αγοράστηκαν εκτυπωτές γιατί για εξωτερικές μελέτες αγοράζουμε εμείς ε, εκτυπωτές, δεν κατάλαβα. Επίσης αυτή τη γενική εικόνα της Γενικής Διεύθυνσης ε, Επικοινωνίας υπάρχουν και ε, ε, πολυθρόνες οικαία, ε, δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό. Και άλλος εξοπλισμός, 71.000 ευρώ, δεν κατάλαβα, από πού προέρχονται όλα αυτά. Και μετά υπάρχουν ορισμένε εταιρείε οι οποίε πραγματικά πληρώθηκαν πολύ χοντρά. Ισάκο Μπέρζον, 22 εκατομμύρια ευρώ και μετά αναρωτιέμαι τι κάνει η Γενική Διεύθυνση της Επεξεργασίας Δεδομένων που έχει ήδη 158 εκατομμύρια ευρώ εάν όλα όσα πρέπει να κάνει τα αναθέτει σε εξωτερικές υπηρεσίες. Ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία δηλαδή που τις δίνουν αυτές οι εξωτερικές συμβουλευτικές εταιρείε για να πληρώσει τόσα πολλά χρήματα. Θα ήμουν ευτυχής με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Και αν δεν πάρουμε τις απαντήσεις έχουμε αυτό πάλι όπως πάντα. Ε, δηλαδή εξω... υπηρεσία ελέγχου του προπολογισμού, διαδικασία του προπολογισμού, επίτροπος κλπ. Ευχαριστώ, Καρλ Χάλτλοντ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για τη μεταφορά 24 που αφορά τη Βαλτική θάλασσα. Κατανοώ ότι η ευθόρμητη προσέγγιση του Λάσλο ήρθε λίγο καθυστερημένα, αλλά το θέμα αυτό το είχα ξεκινήσει εγώ. Θεωρώ ότι η μεταφορά αυτή συνάδει με τα όσα είχαμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με χαροποιεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδρασε κατόπιν πολιτικής παρακίνησης του Κοινοβουλίου και για μένα η μεταφορά αυτή είναι καθόλου αποδεκτή. Είμαι υπέρ του να την ψηφίσουμε σήμερα, αλλά βέβαια ο εισηγητή θα αποφασίσει και σέβομαι την ε, βούλησή του. Θεωρώ όμω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταφορά. Για να δώσουμε τώρα στην Κομισιόν τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήσει τη κυρία Γκρέσλε και μετά ο εισηγητή θα μα δώσει ε, τι άλλε πληροφορίε που ζητήσατε. Oui, merci, euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην φάση αυτή δεν μπορώ να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλε για τους εκτύπωτες. Αλλά θα το εξετάσω το θέμα. Είμαι στη διάθεσή σας γενικά για να σας μεταφέρω νέες πληροφορίες ε, χωρίς καθυστέρηση. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο το θέμα. Είμαι δε πεπισμένος ότι η τεκμηρίωση θα είναι αποδεκτή. Είναι βέβαια σαφές για μας να υπάρξει μια προσωρινή, μια μερική άρση από το αποθεματικό που να αφορά τα 3.700.000. Και αυτό γιατί έχουμε σεβαστεί την υποχρέωση η οποία μας είχε επιβληθεί εν τω μεταξύ. Και νομίζω ότι όλα τα στοιχεία πλέον είναι διαθέσιμα. Από την άλλη η απουσία αυτή πιστώσεων μας δημιουργεί προβλήματα για να προσλάβουμε παρόχους υπηρεσιών στα πλαίσια της πληροφορικής. Προσπαθούμε λοιπόν από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Πληροφορικής να ξεπεράσουμε αυτό το σοβαρό θέμα το οποίο ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υποθέτω όμως ότι αυτή η ενημέρωση θα έρθει σύντομα ούτως ώστε να μην ξαναθέσει, αναγκαστεί να θέσει το θέμα η κυρία Γκρέσλε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προεπιλογισμού. Ο Λάσος Σόγιαν έχει το λόγο. Ε, Ακούγοντας τα σχόλιά σας, κυρία Πρόεδρε, ίσως θα μπορούσα να προτείνω ότι το υπερψηφίσουμε τώρα. Ελοχεύει πάντα ένας κίνδυνος όμως όταν δίνουμε πολύ αναλυτικές επεξηγήσεις διότι πάντα δημιουργούνται νέα ερωτηματικά. Ήταν πλήρως κατανόητη η ερώτηση της ΣΥΝΚΕ και η απάντηση μέχρι τώρα που λαμβάνουμε είναι μια υπόσχεση ότι θα μας απαντήσουν. Το ερώτημα είναι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει μία απάντηση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση και η καθυστέρηση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση θα είναι επιζήμια, διότι μας είπαν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Και όταν λάβουμε την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας κάνω την τελική μου πρόταση. Ε, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Γενική Διευθυντά, ακούσατε τις απαιτήσεις του εισηγητή. Θα μπορούσατε να απαντήσετε στην ερώτηση του που να μας κάνει κάποια σύσταση. Euh, ναι, Πρόεδρε. Η επόμενη συνεδρίασή σα είναι την 13η και 14η Ιουλίου. Λίγο πριν τις διακοπές δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι για την υπογραφή των συμβάσεων ε, θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο και όλα κινδυνεύουν να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο. Αν ψηφίζετε σήμερα, στην ουσία θα χάσουμε τρεις μήνες. Και όπως σας είπα, είναι επίγον το θέμα από πλευρά των υπηρεσιών τεχνικής, πληροφορικής και ανθρωπίνων πόρων. Νομίζω ότι με ικανοποιητικό τρόπο δώσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένες απαντήσεις στα θέματα των μελετών που έχουν γίνει από εξωτερικούς παρόχους, είτε εταιρείε είτε φυσικά πρόσωπα. Αποδείξαμε ότι είμαστε απόλυτα διαθέσιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και αναλαμβάνω την υποχρέωση ότι θα σας δοθούν όλες αυτές οι υποχρεώσεις στα θέματα τα οποία έχει θέσει η κυρία Γκρέσλε και επιθυμία μου θα ήταν αν είναι δυνατόν να κλείσουμε το θέμα αυτό γρήγορα. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, ε, εξαρτάται κυρίως από σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενική Διευθυντά. Οι κανόνε εμάς για την αντιμετώπιση των μεταφορών υποστηρίζουν την επιθυμία σας να αποφασίσουμε σήμερα, γιατί η δική μας προθεσμία είναι 2 εβδόμου. Και μια που πριν δεν έχουμε άλλη ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας, θα πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα. Είμαι εισηγητής. Άκουσα την απάντηση και δεδομένης κατάστασης προτείνω να υποστηρίξουμε την πρόταση λαμβάνω υπόψη και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν και θεωρώ ότι η πρότασή του είναι ικανοποιητική. Βέβαια, η Κομισιόν θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν η απάντηση δεν είναι σαφής και υπάρχουν προβλήματα, τότε θα υπάρξουν συνέπειε. Βέβαια, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, δεν αφορά τη μεταφορά αυτή και επομένως ε, κάνω θετική πρόταση για τη μεταφορά αυτή. Θα ήθελα να σχολιάσω και τη θέση των συναδέλφων φιλελευθέρων. Όπως είπα και στην αρχή, δεν είχα τη δυνατότητα να συζητήσω με τις άλλες πολιτικές ομάδες, κυρίως με τους φιλελευθέρους, που ήταν οι πρωτοπόροι στο θέμα αυτό. Με την υποστήριξη φυσικά και των άλλων ομάδων για τη στρατηγική. Κατ' εμέ είναι πολύ σημαντική η θέση αυτή και επειδή αυτή ήταν η θέση και της δικής μου πολιτικής ομάδος, εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις από τις υπόλοιπες ομάδες, θα μπορούσα να προτείνω να δεχτούμε και τη λύση της Βαλτικής θάλασσας τώρα. wir jetzt, ähm, Ωραία. Θα ψηφίσουμε τώρα. Ξεχωριστά για κάθε μία. Ποιο συμφωνεί με τον εισηγητή και είναι υπέρ της μεταφοράς 16. Dankeschön. Ευχαριστώ. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Μία αποχή. Ωραία. Μεταφορά υπαριθμών 17. Υπέρ. Κατά. Κανείς. Αποχές μια εποχη αποχή. 19-23 θα τα εξετάσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Και τώρα περνάμε στη μεταφορά υπερθμών 24. Ποιος είναι υπέρ της 24. Ποιος είναι κατά αποχές. Κανένας. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Ομόφωνα αποφασίζεται. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό με την προβλήμα της Επιτροπής και παίρνουμε σημείο 21 που πρόκειται για τα λοιπά τμήματα. Βλάντιμιρ Μάνκα είναι ο εισηγητής. Έχουμε την μεταφορά 02 καταρχήν. Και το δικαστήριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όντω η μεταφορά 2 είναι η μόνη που έχετε στον κατάλογο, αλλά στο μεταξύ έγιναν και κάποιε άλλε μεταφορέ. Έχει, άλλε μεταφορέ. Σε αυτή τη συγκεκριμένη μεταφορά έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα θυμάστε ότι όταν ετοιμάζαμε τον προπολογισμό για το 2010 είχαμε μία ενιαία οριζόντια τροπολογία όπου όλα τα θεσμικά όργανα που είχαν δική τους, δικό τους τμήμα μετάφρασης Ε, είχαν ένα αποθεματικό, αλλά αν υπήρξε συνεργασία μεταξύ των θα μπορούσε να διαγραφεί αυτό το ποσό. Το 2006 το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του είχε διαπιστώσει ότι όταν φτάνουν τα διάφορα όργανα στο τέλος των ε, ε, προπολογισμών τους, έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, την δική τους υπηρεσία μετάφρασης, ε, προσλαμβάνουν εξωτερικούς μεταφραστές χωρίς να ελέγξουν αν υπάρχουν ε, δυνατότητες μετάφρασης από άλλα όργανα. Και έτσι χάθηκαν το 2006 περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μας λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Ζητήθηκε λοιπόν από όλα τα θεσμικά όργανα να αποδείξουν ότι χρησιμοποιούν τον προπολογισμό τους για τη μετάφραση και μετά ελέγχουν αν λειτουργούν οι άλλες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο είναι σημαντικό γιατί το δικαστήριο χρειάζεται νομικούς μεταφραστές, είναι πιο εξειδικευμένη η μετάφραση και το δικαστήριο έχει μεγάλο φόρτο εργασίας σε θέματα μετάφρασης, γι' αυτό και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει άνω του 43% τον Ιούλιο των δυνατοτήτων του. Το άρθρος εργασίας ήταν τεράστιο και οι μεταφραστές στο δικαστήριο δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να εργαστούν για άλλα θεσμικά όργανα. Προτείνω λοιπόν να δεχτούμε την αποδέσμευση του αποθεματικού ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. E, και νομίζω ότι μπορούμε να το ψηφίσουμε από εκεί πέρα. E, e, Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο βέβαια το οποίο υπάρχει για σχεδόν όλα τα θεσμικά όργανα. Στο μέλλον δηλαδή θα τα χρησιμοποιούμε ως πακέτο. Δεδομένου όμως ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέθεσε έγκαιρα την αίτησή του και επειδή είναι μια ειδική περίσταση, προτείνω να δεχτούμε αυτό το μεμονωμένο περιστατικό και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα να τα εξετάζουμε ως ε, δέσμοι κονδυλίων. Yeah. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eh, Eh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω μήπως πρέπει να αντικαταστήσουμε τον όρο μεταφορά με τον όρο βυρμά στα, γαλλικά. Αναφέρεστε στο C4. Συγγνώμη, σας διακόψω. Ίσως δεν είναι σαφής προηγουμένως. Υπάρχει μια δέσμη πάνω στην οποία μίλησε ο Βλαντιμίρ Μάνκα τώρα. Πρόκειται για πόρους για μετάφραση και για την Οικονομική ε, ε, Επιτροπή, το Δικαστήριο, την Κομισιόν, όλα μαζί, όλα μαζί. Και ακριβώς ο Βλαντιμίρ Μάνκα μας είπε ότι θα πρέπει να τα εξετάσουμε και ως δέσμοι. Αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να αφαιρέσουμε τίποτα και αν εσείς τώρα το συζητάτε, και λέτε ότι υπάρχουν μεταφορά για το κοινοβούλιο εδώ, αυτό είναι στο δεύτερο τμήμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο θα αφήσουμε τη δέσμη αυτή ενωμένη ή εάν θα αφαιρέσουμε ένα τμήμα όπως προτείνει ο εισηγητής. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτική όταν εξετάζω το θέμα της αφαίρεσης κάποιων συγκεκριμένων θεμάτων γιατί νομίζω ότι ε, προχωράμε πολύ καλύτερα εάν όλες τις οργανώσεις έχουμε σε μία μεταφορά. Θα πρέπει να το σκεφτούμε. Με συγχωρείτε που σας διάκοψα, αλλά θα φτάσουμε σε αυτό που θέλετε να πείτε σε λίγο. Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για ένα ενίο πακέτο. Υπήρξε όμως μία πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε γέρος και για μένα πρόκειται για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, διότι υπάρχουν γλωσσομαθείς νομικοί και πραγματικά υπάρχουν πολλά κατεπήγοντα θέματα, τα οποία απαιτούν ε, πολύ ταχύτατη ψηφοφορία του θέματος αυτού. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα δούμε ως ένα ενιαίο πακέτο, στη διάρκεια τη εβδομάδα θα ακούσουμε και μία ανάλυση για το σύστημα μετάφρασης και θα ήθελα να περιμένω το αποτέλεσμα αυτής της αναλύσεως και κατόπιν να δούμε τι θα γίνει. Θα ήθελα λοιπόν να ψηφίσουμε τα υπόλοιπα σημεία στην επόμενη συνεδρίαση. Για το δικαστήριο όμως θα ήθελα να προτείνω να ψηφίσουμε σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε άλλο. Συμφωνούμε με την πρόταση. Ωραία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν. Ποιος συμφωνεί με τη μεταφορά για τους ε, νομαθείς γλωσσολόγους να σήκω το χέρι του παρακαλώ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Κανένας. Ομόφωνα λοιπόν. Πολύ ωραία. Τα άλλα τμήματα της δέσμης παραμένουν και θα τα εξετάσουμε στην επόμενη μας συνεδρίαση. Και ψηφίζουμε στους κολλούς. Τώρα περνάμε στις μεμονωμένες μεταφορές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλαντιμίρ. Ναι. Να ξεκινήσουμε με το C5. Προσωρινός απασχολούμενο προσωπικό. Ε, να υπενθυμίσω ότι είμαστε στα τέλη Ιουνίου, έχουμε γκρίνει κάποιες τροποποίησεις ε, προς την κατεύθυνση της συνθήκης Λισαβόνα. Τώρα εδώ τι θέλουμε να κάνουμε. θα πρέπει με αυτό το προσωπικό να έχουμε τη δυνατότητα να γίνουν τα όσα είναι απαραίτητα για τις αλλαγές και τις μετατροπές βάσει της συνθήκης Λισαβόνας. Αν χρειαστεί θα γίνουν διαγωνισμοί για προσλήψεις προσωπικού, ε, αλλά έχουν ε, εγκριθεί κάποιες θέσεις τέλη Μαΐου και για να γίνει ο διαγωνισμός ενδιάμεσα θα χρειαστεί ένα διάστημα 8 μηνών. Χρειάζεται λοιπόν πρόσληψη προσωπικού ε, για αυτό το διάμεσο διάστημα και οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να προσπαθήσουν να προσλάβουν προσωπικό και να υπενθυμίσουν ότι πρόκειται για προσωρινή ε, ε σύμβαση και όχι μόνιμη σύμβαση προσωπικό. Θέλει κάποιο το λόγο από αυτόν. Όχι. Ωραία. Ποιος θέλει να ακολουθήσει την πρόταση του συγκεκριμένου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Κανένα. Οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Επόμενο σημείο. Για το C1. εργαζόμενοι που σχετίζονται με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς την Κροατία. 150.000 ευρώ πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο από πολιτική σκοπιά, επομένως θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτή τη μεταφορά. Αυτή είναι η πρότασή μας. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με τη μεταφορά αλλά θα θέλαμε να γίνει αφού βεβαιωθούμε ότι η Κροατία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν να προσληφθεί αυτό το προσωπικό αφού είμαστε βέβαιοι ότι θα ενταχθεί η Κροατία. Γνωρίζουμε βέβαια ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος προετοιμασίας, αλλά με αυτή την επιφύλαξη ε, θα εγκρίνουμε την ε, μεταφορά αυτή. Ευχαριστώ. Ich bin nicht sicher, dass wir äh, diese... Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο μπορούμε να επιβάλλουμε την επιφύλαξη αυτή. Παρόλο που οι συνάδελφοι είναι σίγουροι ότι κάποια στιγμή η Κροατία θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι να σας πω. Χρειαζόμαστε βέβαια χρόνο προετοιμασίας για τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να εντάξουν τους νέους συναδέλφους. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε έτσι αυστηρά περιοριστικοί, φοβούμε. Ποιος είναι υπέρ της πρώτης του εισηγητή. Κατά. Αποχές. Ομόφωνα εγκρίνεται. Το επόμενο, δηλαδή, παρακαλώ. Λοιπόν, 22, μεταφορά 22, C3. Μιλάμε για αποδέσμευση αποθεματικών κατόπιν ετήσεως του ΕΛΚ. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αν θέλουν να πούν κάτι, αν συμφωνούν, εμείς μπορούμε να το αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ. οι πληροφορίες που μας έδωσαν για το διαχωρισμό μεταξύ πάγιων και μεταβλητών ε, δαπανών για να είναι μεγαλύτερη η διαφάνεια και να είναι πιο σαφή τα πράγματα ε, είναι επαρκής. Θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε βέβαια, αλλά θεωρούμε ότι αρκούν αυτές οι πληροφορίες και μπορούμε να προχωρήσουμε ε, βέβαια στη διαδικασία ε, υλοποίηση και των άλλων μέτρων ώστε να δικαιολογούνται όλες οι υπόλοιπες δαπάνες. Καλό θα ήταν να προβλέπουμε και λίγα πράγματα γι' αυτό το μεταβλητε, μεταβλητές δαπάνες στο μέλλον. Είμαστε υπέρ όμως της έγκρισης αυτής της μεταφοράς. Derek. Yes, yeah, I would... Ο Ναι κύριε Πρόεδρε. Θα το υποστηρίξω αλλά όπως και ο συνάδελφος ζητήσαμε αυτή το καταμερισμό πάγιων και μεταβλητών δαπανών και λάβαμε και μια ανάλυση πριν από λίγο καιρό. Τα χρειαζόμασταν αυτά για να δούμε πού ξοδεύουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Ε, θεωρώ ότι αυτό είναι πιο σημαντικό. Καλό θα ήταν βέβαια να κάνουμε και μία συζήτηση για να δούμε τι γίνεται στο μέλλον με αυτές τις πάγιες και τις μεταβλητές δαπάνες για να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η επόμενη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει εδώ στην Επιτροπή μας. Gut, Dank. ευχαριστώ. Ποιος ακολουθεί την πρόταση του συζητή. Κατά. Ωραία. Ε, ομόφωνα είναι κρίθη. Τελευταία μεταφορά. Οκ. Okay. Ε, πρώτος υπεριθμών 2. Διορθωτικός προπολογισμό 02, Επιτροπή των Περιφερειών και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή η μεταφορά και προκύπτει επειδή αλλάζει ο τίτλος της συνθήκης της Λισαβόνας. Κυρία Πρόεδρε, προς το παρόν δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. συζητάμε στις τριμερείς συνομιλίες της 30 Ιουνίου, διότι πραγματικά είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να επιλύσουμε τα πράγματα και θα ήθελα λοιπόν όλοι να εγγράψουμε το σημείο αυτό στις τριμερείς συνομιλίες που θα έχουμε στις 30 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο εισηγητής είναι ο συμπραγματικός διορθωτικός προϋπολογισμός υπ. 2 που ξέρουμε ότι εξετάζεται και στο Συμβούλιο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι κάτι που έχουν οι συνάδελφοι στο φάκελό τους, που τον έλαβαν από τη γραμματεία. Πρώτα για μία μεταφορά 20.000 ευρώ. Υπερψηφίζουμε ή όχι. Η μεταφορά αυτή αφορά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 20.000 ευρώ για ε, δικαστικές δαπάνες. Τεχνική προσαρμογή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα υπερψηφίσουμε. Ποιος θέλει να ακολουθήσει τον εισηγητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Κανένας. Αποχές. Επάλλη κανένας. Ωραία. εκμεταλλευτήκαμε καλά λοιπόν τον χρόνο ψηφοφορία που είχαμε. Και μια που εξακολουθώ να μην βλέπω τον Ρομπέρτο Γιαλτέρη που θέλει να μας κάνει μια παρουσίαση για τη χθεσινή συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Επιτροπής και της Σύμπαντης Εκπροσώπου και του Κοινοβουλίου. Θα εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας και θα σας πω τι αποφάσισαν οι συγγητές χθες και ποιες είναι οι προτάσεις που κάνουν. Και όποιος διαφωνεί, παρακαλώ να πάρει το λόγο. Πρώτον, σταθερικός προπολογισμό ως υπαριθμών 5. Εισηγητής Λάσλο Σόγιαν. Σταθερικός προπολογισμό υπαριθμών 6. δεν προτρέχουμε νομίζω, λέγοντας ότι αυτό θα πρέπει να τεθεί στα λεγόμενες άλλες υπηρεσίες. Ο Βλάντιμιρ ε, Μάνκα και ο Λάσλο λόγιαν είναι λοιπόν εδώ ε, συνεισηγητές. Στο σημείο 3 οι εισηγητές αποφάσισαν να με στείλουν αύριο στην Πάρμα, μια που είμαι μόνιμη εισηγήτρια για τις εξωτερικές υπηρεσίες, μαζί με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και βέβαια θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα κατόπιν. Η ομάδα των σοσιαλιστών θα αναλάβει την γνωμοδότηση για την έκθεση της Επιτροπής Έρευνας και Βιομηχανίας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχετικά σχέδια. Πέμπτον, συμφωνήσαμε να κρίνουμε την γνωμοδότηση Καλτιέρη στην επόμενη συνεδρίαση, βέβαια μέσα στα πλαίσια για του χρονοδιαγράμματος. που ορίστηκε από την ΑΦΕΤ και πάντα σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η χθεσινή συμφωνία. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε συμφωνία, θα το δούμε βέβαια. Έκτον. Συζητήσαμε πώς οι με εφαρμοστικών μέτρων, τα μέτρα που χρειάζονται δηλαδή ουτω ώστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερικη Δράση να εγκαθιδρυθεί και να αρχίσει να λειτουργεί ω τεχνικέ δηλαδή προποθέσει, θεωρούμε ότι το πρώτο τμήμα θα υιοθετηθεί στη δεύτερη σύνοδο του Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο και ο διορθωτικό και στην πραγματικό προπολογισμό υπαριθμών 6 που είναι εισηγητέ Σούριαν Μάνκα θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί σωστά για να μπορέσει να ενταχθεί σε όλες αυτές τις απαιτήσει. Έβδομο. Συζητήσαμε πώς οι επιπτώσεις της συνθήκης Λισαβόνας και η προσαρμογή τους στους διάφορους κανόνες που έχουμε εμείς για τη λειτουργία μας θα πραγματοποιηθεί. Δηλαδή και τον δημοσιονομικό κανονισμό και την MFF. Και τη νέα πρόταση για την διαθεσμική συμφωνία όλα αυτά θα τα εξετάσουμε σαν δέσμη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε όλα αυτά με τη σειρά. Καταρχήν, να προσαρμόσουμε τον δημοσιονομικό κανονισμό για τις ε, υπηρεσίες εξωτερικής δράσης Ανάφερε η κυρία Κρέσλε ότι το θέμα του άρθρου 1 παραδείγματο χάρη καταρχήν θα αναφέρεται μόνο στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης μετά και στα άλλα όργανα. Δεύτερον, δεν θεωρούμε ότι αν μπορώ να το πω η δέσμη της Λιζαβόνας θα πρέπει να ανοίξει γιατί ξέρουμε ότι και η μεσοπρόθεσμη μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός κανονισμός και οργάνωση χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ε, μια διαδικασία συναπόφασης τόσο ώστε να μην η δέσμη αυτή ενωμένη και να έχουμε δυνατότητα να την επιβάλλουμε. Οι συντονιστέ προτείνουν λοιπόν αυτή η δέσμη Λισαβόνα να μην ανοίξει, να μείνει έτσι όσο έχει, δεμένη. Ούτω ώστε ενδεχομένω αυτό που είπε προηγουμένως η Ίγκεμποργκ, για το θέμα της τριετούς αναθεώρησης. Αυτό θα πρέπει ή να ενταχθεί ή να περάσει το δεύτερο τμήμα. Αυτές είναι οι προτάσεις των συντονιστών όπως του χθε το βράδυ. Εάν διαφωνεί κάποιος πρέπει να διαφωνήσει τώρα, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι αποφασίστηκε. Ίγκεμπαρκ. Δεν θέλω να επανέλθω στη συζήτηση που είχαμε. Συμφωνώ με την άποψη αυτή. Αυτό το είχαμε πάντα κατά νου όσον αφορά τη Λισαβόνα και το δημοσιονομικό κανονισμό. Αλλά ακριβώ αυτή η μεταρρύθμιση, η επαναδιατύπωση είναι το πρόβλημα. Και όπως είπε και ο Ράνερ, θα ήταν καλά ο δημοσιονομικός κανονισμός να ακολουθήσει τον άλλον για να μπορέσουμε να διακανονίσουμε όσα δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Εφόσον δεν έχει λυθεί το θέμα λοιπόν της διατύπωσης, θα πρέπει να παραμείνουμε επιφυλακτικοί. Ευχαριστώ. Δεν έχω κάποιο σχόλιο γι' αυτό, ένα άλλο σχόλιο σχετικά με το 6. Εμείς είπαμε ότι θα θέλαμε να αντικαταστήσουμε τον κύριο Μάνκα με τον κύριο Γκαλτιέρη που ήταν υπεύθυνο για την εξωτερική υπηρεσία. Αλλά δεν έχουμε πάρει την τελική απόφαση, θα ήθελα ίσως όμως να αλλάξουμε τον εισηγητή. Εγώ είμαι συνεισηγητής. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουμε επίσημα στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Ναι. Ναι, να το αφήσουμε αυτό. Είναι η επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών των ε, συντονιστών. Και το σύστημα τότε. Είναι πάντα προβληματιστικό κατά τη γνώμη να κάνουμε κάποιες αλλαγέ έτσι ξαφνικά. Γιατί ήδη το θεώρησα πολύ προβληματικό ότι το ΕΛ ξαφνικά μας έδωσε άλλο εισηγητή αντί το Ράμε για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Δεν διαφωνώ με το συνάδελφο που ορίστηκε, αλλά είμαι κατά του να κάνουμε αυτά τα πράγματα έτσι ξαφνικά, να κάνουμε έτσι ε, κάποιες κινήσεις νευρικές ε, και αν στραφώ προς τον ΕΛΚΑ ε, ε, βλέπω ότι ο Σαλβαδό δεν έχει καμία αντίληση. Τέλο πάντων, θα το δούμε την επόμενη φορά στη συνεδρίαση των συντονιστών. Zu Ingeborg, Ingeborg, ich verstehe das. Ingeborg, ε, καταλαβαίνω αυτά που είπες. Αλλά χρειάζομαι χρειάζομαστε τώρα το δικό μας δημοσιονομικό κανονισμό για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια μέσα στα χέρια μας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το φάκελο του Ράιμερ. Μα δεν υπάρχει αντίφαση. Ναι, ναι. Θέλω να είναι σαφές ότι υπάρχει κάποιος λόγος γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Dann schließen wir das ab. Ωραία, μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το σημείο. Βλέπω, ακόμα δεν έχει έρθει ο εισηγητής μας. Νομίζω ότι είναι στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ωραία. Περάσουμε στο σημείο 15. Συμφωνία Ελευτική Σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νήσων του Σολομόντος. Πρέπει να εγκρίνουμε σε μια συμφωνία αλλιευτική με, τα νησιά του Σολομόντος. Είναι πολύ μικρή η συμφωνία αυτή, ίσως είναι η πιο μικρή από όλες τις αντίστοιχες. Και τα Solomon Islands Ξέρετε ότι δεν είναι και ιδιαίτερα ανησυχητικέ χώρες, ούτε χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ε, διαφθορά, δεν υπάρχει θέμα λοιπόν. Κάποιε σκέψεις όμως είναι απαραίτητες. Πρώτον, ότι το 2010 στην ουσία μας ζήτησε τον Απρίλιο του 2010 να βγάλουμε μία γνωμοδότηση για μία απόφαση του Συμβουλίου η οποία είχε εκδοθεί το 2009. Αυτό τώρα το εκ των υστέρων είναι λίγο μυστήριο. Αλλά εν πάση περιπτώσει η συμφωνία αυτή έγινε σε μια κεντρική κομβική περίοδο και δεν θα πρέπει να τον μπλοκάρουμε σε επίπεδο διαδικαστικό. Εμείς θα πρέπει επίσης να συνοδεύσουμε τις, ε, την απόφασή μας από κάποιες ε, γενικότερες σκέψεις που θα έλεγαν κυρίως, περιγράφουν κυρίως την επιθυμία μας να προστατεύονται ε, τα, τα αλλιεύματα τα οποία αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στις τοπικές αλλιευτικές δραστηριότητες, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα Salomon Islands. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ. Παρατηρήσεις από αυτού. Η κυρία Δουλό, όχι. Ποιος. Α, παρακαλώ. Εστέλ. je, vois que la Η αλία δεν συγκίνει πάρα πολύ κόσμο στην επιτροπή αυτή, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτά που έλεγε ο Αλφονσί και να πω ότι η διαδικασία αυτή είναι λίγο διφορούμενη. Ζητάνε τη γνώμη μας 7 ε, μήνες αργότερα και αυτό είναι λίγο θα έλεγα περίεργο αν μη τι άλλο. Αλλά για να δούμε ακριβώς τι προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, είναι σαφές ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η μέθοδος εργασίας στην οποία χρησιμοποιούν τα όργανα. Θα πρέπει επίσης η Επιτροπή Αλληλείας, η οποία είναι επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή, να εκφέρει τη γνώμη της, γιατί α, αλλιώς δεν θα μπορούμε ούτε κι εμείς να εκφέρουμε τη δική μας νομοδότηση. Και αυτό είναι σοβαρό θέμα, γιατί ξέρετε ότι οι διεθνείς αλληλευτικές συμφωνίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της ε, πολιτικής, της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και να πω επίσης ότι η συμφωνία αυτή αντιπροσωπεύει περίπου 400 εκατομμύρια κατέτος, αλλά έρχεται μια αντίστοιχη συμφωνία με τη Μαυριτανία, η οποία ε, φτάνει στα 3 εκατομμύρια κατέτος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα. Όλοι λέμε ότι η διαδικασία της Λισαβόνας είναι εξαιρετική και βελτιώνει τις διαδικασίες, αλλά βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο θεωρητικά μόνο έχει περισσότερες αρμοδιότητες ε, από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να οργανωθούμε καλά. Και σχετικά με την αρχική συμφωνία, τα θέματα αλληλείας έχουν, ε, θα έλεγα, σχετικά χάσει λίγο τη σημασία τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε ο εισηγητής, σε αυτή τη φάση της συμφωνίας με τα Solomon Islands προσπαθούμε να ορίσουμε σωστά την θέση σε λειτουργία, σε ισχύ θα έλεγα, της συνθήκης της Λισαβόνας. είναι σαφές ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παλές διαδικασίες χωρίς να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να ζητείτε η γνώμη μας στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης με έξι μήνες διαφορά. Τελειώνω λέγοντας ότι ας πούμε ότι είναι τυχαίο το συγκεκριμένο συμβάν. αλλά πρέπει να το υπογραμμίσουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε οι συμφωνίες οι αλλιευτικές να υπογράφονται έγκαιρα και να μην ζητείται η άποψή μας μόνο εκ των υστέρων. Σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας με τα νησιά Σολομόντος. Στην ουσία θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το οποίο ίσχυε τα προηγούμενα τρία χρόνια με την χώρα αυτή και δεν έχουμε καμία διαφορά ούτε δημοσιονομική ούτε σε επίπεδο δαπανών γενικότερα. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, η μόνη φορά που είχαμε κάποιο πρόβλημα με την Επιτροπή Αλίας για την υπογραφή και χρηματοδότηση αλληλευτικών συμφωνιών ήταν ε, το 2000 τότε που ε, ανανεώθηκε η Συμφωνία Λία με το Μαρόκο. Βέβαια, σαφώς οι ποσότητες για τις οποίες μιλούσαμε τότε ήταν πολύ υψηλότερες από αυτές που έχουμε σήμερα. Αλλά από την άλλη, η συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί ένα νέο σύστημα ε, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αλλίας μπορεί να έχει περισσότερη επιρροή σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες. Επομένως, αλλάζουν η ε, ισορροπία σχέσεων μεταξύ Επιτροπής Αλίας και Επιτροπής Προϋπολογισμού στο μέλλον. Πρότασή μου, κυρία Πρόεδρε, είναι να προσκαλέσουμε κάποιον από την Επιτροπή Αλίας, ε, την Πρόεδρο ή κάποιον από το Προεδρείο, στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμού, δεν ξέρω αν θα γίνει τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο, για να υπάρχει ένας τρόπος ε, συνεργασίας για το μέλλον, ώστε να μην έρχονται αυτές οι αιτήσει χρηματοδότησης ε, συμφωνιών αλίας καθυστερημένα. Ε, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εργασία αυτή, διότι θα καθορίσουμε και τους κανόνες λειτουργίας για το μέλλον. Πολύ καλή αυτή η ιδέα σας. Το Ιούλιο ίσως δεν προφτάρουμε. Σεπτέμβριο όμως θα μπορούσαμε πραγματικά να προβλέψουμε κάτι τέτοιο για συνεργασία με την Επιτροπή Αλληλείας. Γιατί συνήθως μείνουν, μένουν εκτός ε, νηφώνους και η Επιτροπή Προϋπολογισμού και η Επιτροπή Ελίας. Και η Κομισιόν κάνει τι θέλει. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Όχι. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι. Από ό,τι μου είπανε δεν χρειάζεται γιατί ο, η Κάτια είπε ότι αυτή η επιτροπή την οποία θα έπρεπε να ενημερώσω για την προσπάθεια που καταβάλει το ε, Κοινοβούλιο για την ισότητα είναι βέβαια, θα παραμείνω εδώ, είναι βέβαια κάπως περίεργο γιατί ούτε ο πρόεδρος είναι παρόν αλλά και οι τρεις αντιπρόεδροι επίσης λείπουν. Λοιπόν, περνάμε τώρα. Πού είναι ο Ρομπέρτο, μόλις τον είδα. Α, εκεί. Άρε, Ρομπέρτο. Θα μας πει ο Ρομπέρτο τι έγινε χθε στη Μαδρίτη και τι συμφωνήθηκε επίσης. Παρακαλώ, Ρομπέρτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω ένα πρώτο έγγραφο και να σας παρουσιάσω επίσης προφορικά και το τι έγινε στη χθεσινή συνάντηση στη Μαδρίτη. Το έγγραφο αυτό, το οποίο δεν είναι το τελικό επίσημο έγγραφο και σίγουρα θα έχει κάποια επιμέρους τεχνικά στοιχεία, λεπτομέρειες προς διόρθωση, η γνωμοδότησή μου αυτή στην έκθεση Μπροκ Verhofstadt διαφέρει από το κείμενο εργασίας πάνω στο οποίο κάναμε την προηγούμενη συζήτησή μας και συγκεντρώνει θα έλεγα τα αποτελέσματα της συμβιβαστικής ε, λύσης την οποία κατέληξαν χτες στη Μαδρίτη στα πλαίσια του τετραμερούς διαλόγου του τελευταίου από μια μεγάλη σειρά αντίστοιχων τέτοιων συναντήσεων και που οδήγησε σε ουσιαστικές τροποποιήσεις του αρχικού κειμένου που είχε παρουσιαστεί από την κυρία Άστον και είχε προταθεί στο Συμβούλιο στις 25 Μαρτίου. Επέλεξα τη συγκεκριμένη διαδικασία για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος γιατί πρόκειται για μια διαδικασία διαβούλευσης καταρχάς. Και το να παρουσιάσει κανείς ένα διαφορετικό κείμενο θα μπορούσε ίσως να δείξει καλύτερα αυτό το οποίο θα θέλαμε να πετύχουμε, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να πετύχουμε στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Δεύτερον, το κείμενο αυτό περιλαμβάνει και τη συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξαν χθε, που είναι μια καλή συμβιβαστική λύση, πολύ καλύτερη από αυτές τις οποίες, ε, από τις προσδοκίες, εν τις οποίες είχα εγώ. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, αναλέξετε πιο προσεκτικά ε, το χθεσινό κείμενο με την πρόταση του Μαρτίου της Άστον, έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές σε αρκετά σημεία. να προσθέσω εδώ και κάτι το οποίο δεν είναι στο κείμενο. Στα δέκα σημεία για την λεγόμενη πολιτική ε, της υπευθενοποίησης ή του accountability το δέκατο σημείο εν πολλής κάνει δεκτό το αίτημα της Επιτροπής μας, ε, την τροποποίηση δηλαδή της Διοργανικής Συμφωνίας για τον προϋπολογισμό στον τομέα της αλίας. Και ταυτόχρονα δέχεται ότι για να υπάρχουν βασικές αυτόνομες γραμμές στον προϋπολογισμό για αυτή την πολιτική. Κάτι το οποίο ε, έρχεται εν πολύ σε αντίθεση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ενώ το τελικό κείμενο και το αποτέλεσμα του τετραμερούς διαλόγου τι δείχνουν. Η συμβιβαστική λύση αφορά το συνδυασμό του διοικητικού προϋπολογισμού με ένα άλλο τμήμα διαφορετικό, το δέκατο τμήμα, είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά θα προτιμούσε να πάει στο τρίτο τμήμα. Παρ' όλα αυτά ο συνδυασμός των δυνάμεων και η νομοθετική διαδικασία κατέστησαν εφικτή την επίτευξη αυτού του βέλτιστου αποτελέσματος. Παρ' όλα αυτά, οι τρόποι με τους οποίους θα εφαρμοστεί αυτή η αυτονομία έχουν αλλάξει εν πολλής. Ο διοικητικός προϋπολογισμός και χωρισμένος περιλαμβάνει και κάποια πλεονεκτήματα σύμφωνα με τη γνώμη του Κοινοβουλίου γιατί η διαδικασία απαλλαγής για αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού δεν θα γίνεται στο εσωτερικό της συνολικής απαλλαγής της Επιτροπής, αλλά ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι υπέκειτο μέχρι τώρα θα έλεγα στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ή είχε συμπεριληφθεί στα πλαίσια της ε, Συμφωνίας Κυρίων, τώρα θα αντιμετωπίζεται πλήρως δημοσιονομικά στα πλαίσια ενός ξεχωριστού τμήματος του προϋπολογισμού του Συμβουλίου. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροποποιήσεις σχετικά με την πρώτη πρόταση της 25ης Μαρτίου, αφορούν θέματα προσωπικού, αφορούν θέματα πολιτικής και κυρίως δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ο σχετικός με τις δημοσιονομικές διαδικασίες. Δεν θα ήθελα τώρα να σας δώσω λεπτομέρειες, μπορείτε να τα διαβάσετε στο έγγραφο και τις προτάσεις τροπολόγησης οι οποίες έχουν γίνει. Γίνονται λοιπόν κάποιες διευκρινήσεις και δίδονται αρκετές εγγυήσει ιδιαίτερα για τη διαδικασία απαλλαγής και δίδεται στο Κοινοβούλιο η απαιτούμενη τεκμηρίωση έτσι ώστε να φέρει εις πέρας ε, την ε, αρμοδιότητά του σαν ε, αρχή επί της απαλλαγής. Επίσης το ίδιο γίνεται και σε σχέση με τις αρμοδιότητες της ΟΛΑΦ Το ίδιο και με τις ελεγκτικές διαδικασίες λέγεται ότι για τις διοικητικές δαπάνες πρέπει να υπάρξει σύνδεση της εσωτερικής ελεγκτικής διαδικασίας με τη γενικότερη ελεγκτική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς να προκαταλαμβάνεται το ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός μπορεί να αποφασίζει ότι η ελεγκτική διαδικασία μπορεί να γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας της Επιτροπής. Πρόκειται για μια τροπολογία η οποία αναφέρεται στο θέμα της συνεργασίας και όχι στην φύση της ελεγκτικής διαδικασίας. Διαγράφει επίσης και η αναφορά στον είπα το εκπρόσωπο ως διατάκτη, απλά εφαρμόζεται ο κανόνας 59 του δημοσιονομικού κανονισμού, γίνεται καλύτερη διευκρίνηση ανάμεσα στις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες, Προβλέπεται επίσης ότι η διαδικασία θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα γενικότερο έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών των σχετικών με την εξωτερική δράση της Ένωσης για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες πολιτικού ελέγχου από πλευράς ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν πάση περιπτώσει αυτό το κομμάτι το οποίο αφορά κυρίως το άρθρο 7 Αυτέτε του προϋπολογισμού φυσικά. Εδώ έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις. Ένα δεύτερο κομμάτι θεμάτων που αφορά την Επιτροπή μας αφορά τη διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων, ιδιαίτερα στα πλαίσια της βοήθειας για την ανάπτυξη. Εδώ ο κίνδυνος είναι να δούμε να αφαιρείται από την Επιτροπή η ευθύνη την οποία έχει σχετικά με τα συγκεκριμένα αυτά μέσα. Εδώ έχουν γίνει οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις θα έλεγα, οι οποίες εν πολλής διασώζουν θα έλεγα την κοινοτική μέθοδο. δίδεται μια θα έλεγα συγκεκριμένη ε, διευκρίνηση σχετικά με την επιρροή του υπάτου εκπροσώπου στο σύνολο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα γίνεται αναφορά στη συνδυασμένη παρέμβαση για τον καθορισμό της πολιτικής αυτής της εξωτερικής. Δίδονται συγκεκριμένες ευθύνες σαν παράδειγμα και στον αρμόδιο επίτροπο για τα θέματα της ανάπτυξης, διευκρινίζονται οι δυνατότητες διαχείρισης από πλευράς του συγκεκριμένου επιτρόπου για την ανάπτυξη δηλαδή των μέσων τα οποία έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση και διευκρινίζεται και αναδιατυπώνεται επίσης η μορφή συνεργασίας ανάμεσα στην προετοιμασία των αποφάσεων των τριών πρώτων φάσεων του κύκλου προγραμματισμού των υπηρεσιών αυτών, της υπηρεσίας αυτής υπό την ευθύνη του Επιτρόπου και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία συνεργάζεται για την προετοιμασία των πολιτικών αποφάσεων και θα έχει τελικά και την πολιτική ευθύνη πέραν της οικονομικής φυσικά ευθύνης ή καλύτερα της δημοσιονομικής ευθύνης. Τέλος, έχει υπάρξει αναφορά και στο 298, ένα πολύ σημαντικό άρθρο, νέο άρθρο, που δεν υπήρχε στις προηγούμενες συνθήκες και καθορίζεται μια πολιτική συναπόφασης για το σύνολο των αποφάσεων που έχουν σχέση με την αυτόνομη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των μέσων και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισάγει μια διαφορετική νομική βάση από το άρθρο 27, ιδιαίτερος χρήσιμη για το μέλλον και για τα, μελλον, τις μελλοντικές φάσεις, εν πάση περιπτώσει, αυτές που θα ακολουθήσουν στο μέλλον την ζωή αυτής της νέας υπηρεσίας. Συνεπώς, εγώ κρίνω με θετικό τρόπο τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από πλευράς χρονικής θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πολιτικά το κοινοβούλιο αυτό να καταφέρει να υιοθετήσει την έκθεση αυτή Μπροκ Φερχόστατ πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω και τους πολιτικούς λόγους οι οποίοι επιβάλλουν αν θέλετε τη συγκεκριμένη επιλογή. Το Συμβούλιο δεν είναι ευχαριστημένο από το αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε καταλήξει. Το Συμβούλιο θεωρούσε ότι δεν είναι τροποποιήσιμο αυτό το οποίο ε, είχε αποφασιστεί στις προηγούμενες συναντήσεις και πιστεύω ότι αν εμείς έχουμε την δυνατότητα της ταχυτά της έγκρισης των δύο νομοθετικών εγγράφων το διοικητικό δηλαδή που αφορά το προσωπικό και τον οικονομικό κανονισμό, τότε δεν θα χρειαστεί να ζητήσουμε περαιτέρω τροποποιήσεις και θα έχουμε την δυνατότητα όχι μόνο απλά να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας στον τομέα των δημοσιονομικών, αλλά θα έχουμε και την δυνατότητα σε εισαγωγικά αντιμέτρων στην περίπτωση που υπάρξει τροποποίηση από πλευρά Συμβουλίου των Συμπεφωνημένων. Συνεπώς, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια γρήγορη σχετικά διαδικασία για την έγκριση των αποτελεσμάτων αυτών και γενικότερα για την σωστή και ευθέτη χρονικά εφαρμογή της εκθέσεως Μπροκ Φερχόστατ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κολτιέρη. Προτείνω αν δεν έχετε αντίρρηση, να περάσουμε στο επόμενο σημείο και να κάνουμε μια συζήτηση μετά και για τις δύο εκθέσεις, γιατί ε, είναι αλληλένδετες. Ναι, ευχαριστώ. Ο δημοσιονομικός κανονισμός στην περίπτωση αυτή ακολουθεί όλο το δικοδόμημα, το σύστημα του ελέγχου από πλευράς Κοινοβουλίου και αν ε, δεν θεωρηθεί ο οργανισμός ε, ανεξάρτητος αυτή η υπηρεσία, ε, δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτό. Σαφώς το Συμβούλιο θα τη στηρίξει αυτές τις τροπολογίες. Πάντα μας έλεγαν ότι θα υπάρχει μια πραγματική συζήτηση. Θα γίνει μια πραγματική συζήτηση. Βέβαια, η αποδοχή από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ καλό που έχουμε τάπητος τώρα αυτά αποτελέσματα, αλλά αυτή η ομάδα δεν είχε καμία εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρχε εντολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Και αυτό τώρα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το αποτέλεσμα, θα το κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα να δώσουμε τη δυνατότητα στις πολιτικές ομάδες να αποφασίσουν τι θα πρέπει να γίνει από εκεί και πέρα και νομίζω ότι θα ήταν καλό να λάβουμε πολύ σοβαρό υπόψη την συναπόφαση. Συναπόφαση σημαίνει ότι πραγματικά συναποφασίζουμε ότι δεν πρέπει να παρακαλάμε. Γιατί έχουμε τη συναπόφαση ε, και σχετικά με το κανονισμό για το προσωπικό και τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Αλλά ό,τι γίνει έγινε. Ό,τι δεν πετύχουμε τώρα δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Και ό,τι πετύχουμε τώρα μέσα στα πλαίσια του ε, κανονισμό του Συμβουλίου μπορεί μετά να ε, καταγγελθεί μονομερός. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε την υπηρεσία αυτή εξωτερικών δράσης να... που έχουμε σε ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό και να δούμε ότι η διαφορές αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κομισιόν και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στις αντιποστολές αυτές να διευκρινιστεί γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε έγινε όλα αυτά που συζητάμε τώρα εδώ και πολύ καιρό είναι θέματα προς απόφαση πια ποτέ δεν απόκρυψα ότι εγώ βλέπω εδώ να υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα και υπάρχει και για την είπα το εκπρόσωπο η οποία ό,τι σφάλμα να γίνει θα βρίσκεται στην πουκά του κανονιού όλου του κόσμου. θα ήταν... Θα έπρεπε ίσως να χαρώ αν θέλει γιατί θα διασκεδάσω τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν είναι αυτό ο στόχος. Και αυτή η ομάδα διαπραγμάτευσης χωρίς εννοή μας είχε υποσχεθεί πάντα ότι δεν είναι δεσμευτικό για κανέναν και μετά θα υπάρχει σωστή διαδικασία διαβούλευσης. Τώρα όμως μας αφαιρείται αυτή η δυνατότητα διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ενισχυτικό γιατί στο τέλος θα υποφέρει η ίδια η υπηρεσία και είμαι πολύ αισιόδοξη ότι το Συμβούλιο χαίρεται ότι το πέτυχε τώρα, αλλά εντάξει, 50 χρόνια δεν το είχαμε, τώρα να το έχουμε ένα μήνα παραπάνω δεν πειράζει. Αλλά θα πρέπει νομίζω να ε, υπάρχει μια ομάδα που θα έχει ευρύτατε αρμοδιότητε, γιατί με την ανάμειξη του εσωτερικού του δημοσιονομικού κανονισμού έχουμε 8 δισεκατομμύρια ευρώ στον ε, λειτουργικό τμήμα. Αν έχουμε λοιπόν εδώ περισσότερο έλεγχο στον προπολογισμό εδώ, <coughs> τη Επιτροπή Εξωτερική Δράση, είναι περισσότερα αυτά που κερδίζουμε από εκείνα που παραδίδουμε. Και θα πρέπει οι δυσκολίες στην διαδικασία απαλλαγής να εξεταστούν, να συζητηθούν και εάν πρόκειται να παραδώσουμε κάποια δικαιώματα, ε, θα μπορούσα να πω παραδείγματος, χάρη και κάτι άλλο, ότι το, η ενσωμάτωση στον ε, προπολογισμό της ε, υπηρεσίας ε, εξωτερικής ενίσχυσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ η υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχει ένα μεικτό χαρακτήρα και ο μεικτός χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και αναφέρομαι εδώ και σε μια γνωμοδότηση της, του Ελεκτρικού συνεδρίου και θα πρέπει νομίζω να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα να αποχωρήσουμε κάποιες αρμοδιότητες ξεκάθαρα και να τις διευκρινίσουμε. Έχω και ένα πρόβλημα με το σημείο 3 και 4. Το συζητήσαμε ήδη το πρωί. Δεν θα πρέπει να περικόψουμε τι αρμοδιότητε των συναδέλφων μέσω τη ε, υπηρεσία εξωτερική δράση. Θα πρέπει να τολμήσουμε, να συζητήσουμε ανοιχτά και τα μειονεκτήματα που δεν βλέπω να υπάρχουν να τα δεχθούμε. Και επίσης ο κύριος Ραπκάε που είναι εισηγητής για τον ε, κανονισμό του προσωπικού συμφωνεί απόλυτα μαζί μας. Πήραμε ένα σχέδιο εδώ, το οποίο δεν έχει και αριθμό μάλιστα. Αυτό το σχέδιο όταν υπάρχει στις διάφορες γλώσσες τότε θα μπορέσουμε μονάχα να ορίσουμε ένα, μια προθεσμία και δεν μπορούμε από τώρα να πούμε αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά τον Ιούλιο ή ε, θα πρέπει να πάμε Σεπτέμβριο και δεν πρέπει να ε, δώσουμε την ύποση ότι αυτό από αυτό θα εξαρτηθεί το μέλλον της ανθρωπότητας, θα πρέπει να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε ανοιχτά με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Κύριε θα ήθελα να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν τέσσερα έγγραφα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το πρώτο είναι το κείμενο του κυρίου Γκουαλτιέρη και βάσει αυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δυνατότητα στην εδώ. Εξ όσων κατανοώ εγώ, η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε χθε ήταν ότι αυτό θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος ε, του καλοκαιριού, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα υπόλοιπα, οι προστίκες στον προπολογισμό, τα θέματα του κανονισμού, θα ψηφιστούν μέχρι το Σεπτέμβριο και από εκεί και πέρα το Κοινοβούλιο έχει κάποιες εξουσίες βάσει διαδικασίας συναπόφασης. Για αυτά τα τρία σκέλη δηλαδή. Πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό των διαδικασιών. Για τα τρία αυτά έγγραφα έχουμε δυνατότητα στην απόφαση, ενώ για το πρώτο δεν έχουμε καμία δυνατότητα στην απόφαση. Η κυρία Τρούπελ. Αδιαδικαστικό, κύριο Σπίγκερ. Για τη συζήτηση που λαμβάνω χώρα αυτή, ποιο αποφάσισε χθε, ποιο. ίσως δεν έγινε κατανοητός, εχθές υπήρξε συμφωνία μεταξύ των συντονιστών της Επιτροπής. Όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση εχθές, αποφάσισαν μια απόφαση που δεν είναι δεσμευτική για το Κοινοβούλιο, έτσι ούτε και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Έχουμε δύο διαδικασίες όμως για τα τέσσερα έγγραφα. Αυτό ήθελα να επισημάνω εγώ, ότι είναι δύο διαφορετικές οι διαδικασίες. Η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρά το γεγονό ότι αυτή δεν ήταν εντολή για όλο το Κοινοβούλιο, αλλά εξ όσων κατανοώ εγώ, υπάρχουν διαφορές ως προς του Κοινοβουλίου, αυτό μας επισημάνεται και μόλις τώρα, και από αυτό που βλέπουμε στο κείμενο είναι ότι έχουμε μια σαφή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο. Πρέπει τώρα βέβαια να συζητηθεί το όλο θέμα, αλλά προσωπικά, ακούγοντας τα όσα είπε ο κύριος Γκουαλτιέρη και διαβάζοντας και το έγγραφο για πρώτη φορά, νομίζω ότι έχουμε επιτύχει κάποια σημεία και έχουν βελτιωθεί κάποια σημεία ε, που αφορούν εμάς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συνδυασμό των συμφερόντων του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα και εκ μέρους ενός μέλους της ε, ΑΦΕΤ και ΕΜΟΥ ως μέλος Επιτροπής εδώ, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκουαλτιέρη το εξή. Ο τρόπος ε, της διαδικασίας που αποφασίστηκε να ακολουθηθεί φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργούνται νέε θέσει μόνο όταν κάποιο κράτο μέλο θέλει να αποστείλει νέα πρόσωπα και όχι όταν εμεί του χρειαζόμαστε ω κοινοβούλιο από πολιτική σκοπιά υπάρχουν 20 αναπληρωτές επικεφαλής αποστολές και 20 ε, υπάλληλοι, τους οποίους θα ήθελαν να καθορίσουν τα κράτη-μέλη. Οι θέσει εργασία θα πρέπει να κατευθύνονται από τις πολιτικές προτεραιότητες, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πολυμερείς θέσει εργασία στο Ηνωμένα Έθνη και όχι μόνο 20, κυρίως για τα θέματα διαχείρισης κρίσεως. Μπορείτε να μας σχολιάσετε, συζητήθηκε το όλο θέμα, το πώς θα γίνει ο καταμορισμός των θέσεων εργασίας και το κατά πόσον θα είναι πολυμερείς αυτές οι θέσεις. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα καλά, ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε εσείς περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Τρούπελ, ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκαλτιέρη και τους άλλους συναδέλφους που πήραν μέρος στην συνάντηση στη Μαδρίτη. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν, αλλά υπάρχει ένα σαφές στρατηγικό θα έλεγα θέμα. Εμείς προσπαθούμε από τη μία να διαπραγματευτούμε τα πάντα και σε μια δεύτερη φάση να καταλήξουμε σε ορισμένες αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η στρατηγική αυτή, όπως είπε, ε, ο κύριος Γουαλτιέρη, είναι να καθορίσουμε ένα πλαίσιο στρατηγικό πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές έτσι ώστε εκ των υστέρων να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει συγκεκριμένες θα έλεγα προτάσεις να κάνει στα πλαίσια της συναπόφασης. Η αίσθησή μου είναι ότι υφιστάμεθα μία κάποια χρονική πίεση προς το παρόν, έντονη και σαν θεσμικό όργανο θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι απαιτείται να υπάρχει ένα πλαίσιο χρονικό μέσα στο οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει τις εργασίες του η εξωτερική υπηρεσία. Υπάρχει ο φόβος ότι θα παραδώσουμε κάποιες δυνατότητες που έχουμε να αποφασίσουμε. Θεωρώ ότι αν κοιτάξουμε το παράμετρο από εκεί από που ξεκινήσαμε, από το, την απόφαση δηλαδή, δηλαδή από το ψήφισμα του Συμβουλίου, πετύχαμε πολύ περισσότερο από εκείνο που μπορούσαμε να περιμένουμε εκ μιας αρχής και νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να εξασφαλίσουμε αυτό που πετύχαμε. Στις διευκρινήσεις που θα υπάρχουν στο οργανισμό του προσωπικού και στον δημοσιονομικό κανονισμό, να τα πραγματοποιούμε θέματα σημαντικά για μας που δεν μπορεί να ορίσει το πλαίσιο αυτό και ταυτόχρονα να φροντίσουμε το Συμβούλιο να τηρήσει αυτά που υποσχέθηκε. Γιατί έχουμε ακόμα αυτά τα όπλα, αν θέλετε, στα χέρια μας. Και έτσι μπορούμε να επιβληθούμε στην συναπόφαση. Κατά τη γνώμη μου, δεν παραδίδουμε καμία δυνατότητα ε, προάσπισης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. των αντίον, μπορούμε να καταδείξουμε ότι τώρα θα πρέπει το Συμβούλιο να κινηθεί προς εμάς, εφόσον εξασφαλίσουμε αυτό που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Ρομπέλτο Γκαλτιέρη. Έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε όλοι νομίζω και αυτόν και τους άλλους διαπραγματευτές της Επιτροπής μας. Έχει συνεργαστεί επίσης στενά με την κυρία Γκρέσλε που έχει και αυτή προσφέρει αρκετά στις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι έχουν ληφθεί όλα αυτά υπόψη σοβαρά. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αρκετές θετικές αλλαγές και σε επίπεδο δημοσιονομικό θα παραμείνουν οι λειτουργικές δαπάνες στο τρίτο τμήμα. Έχουν υπάρξει θετικά βήματα και σχετικά με τη διοργανική συμφωνία, αλλά και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι πετύχαμε αρκετά. Βγάλαμε επίσης τον διοικητικό προϋπολογισμό από τη Συμφωνία των Κυρίων και μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε με τον κανονικό τρόπο. Τώρα για την ύπαρξη ή μη συγκεκριμένης εντολής. σχετικά με τη χθεσινή απόφαση να θυμίσω ότι έχουμε υιοθετήσει μια έκθεση του κυρίου Μπρόκ για την εξωτερική υπηρεσία που καθορίζει τις βασικές γραμμές και πρέπει να γίνουν σεβαστές. Έχουμε δημιουργήσει επίσης μια συγκεκριμένη θα έλεγα προσανατολιστική ομάδα και εκπροσωπούμεθα στη συγκεκριμένη αυτή ομάδα σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στη δική μας πολυομάδα έγινε επίσης και μια συντονιστική ομάδα εργασίας ανάμεσα στους εισηγητές όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών που είχαν εμπλακεί και νομίζω ότι ε, με αυτόν τον τρόπο ορίζουμε σωστά την εντολή προς τους διαπραγματευτές μας. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη εντολή, αλλά είναι σαφές ότι η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο πριν ε, θεωρηθεί έγκυρη. Εγώ έχω έρθει σε επαφή όχι μόνο με την κυβέρνησή μου αλλά και με άλλες χώρες και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πάμε περισσότερο, έστω και λίγο. Εκπλήσωμε που φτάσαμε ως εδώ, γιατί εξ αρχής τα κράτη-μέλη ήταν ιδιαίτερα διστακτικά να δώσουν περαιτέρω αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο ή καλύτερα τα κράτη-μέλη πιέζονται τώρα από την άλλη πλευρά Κάποιες χώρες θεωρούν σαν παράδειγμα ότι η Ισπανική Προεδρία έχει κάνει πιο σημαντικά βήματα από όσο περίμεναν προς την κατεύθυνσή μας. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί λοιπόν σχετικά με τη συμφωνία αυτή και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να σεβαστούμε τη συμφωνία και να υιοθετήσουμε τις βασικές της αρχές το ταχύτερο δυνατόν. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τον Ιούλιο, ελπίζω να μπορεί να γίνει γιατί αλλιώς διατρέχουμε τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα με τα κράτη-μέλη, τα οποία θα μας κατηγορήσουν ότι δεν σεβόμεθα τις ανηλυμένες υποχρεώσεις. Οι λεπτομέρειες σίγουρα θα έρθουν αργότερα, αλλά οι βασικές αρχές θα πρέπει να γίνουν δεκτές το ταχύτερο δυνατόν. Και ναι μεν είμαστε Επιτροπή Προϋπολογισμού και δεν έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά θα πρέπει σαν μέλη αυτού του Κοινοβουλίου να αναλάβουμε τις ευθύνε μας για τη δημιουργία μια σωστής σκέπα και των μέσων που απαιτούνται για να εφαρμοστούν οι αποφάσεις μας και οι διατάξεις της συνθήκης. Ευχαριστώ πολύ. Ο ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή πραγματικά να εξετάσει κανείς όλες τις λεπτομέρειες αυτού του κειμένου. Και ενθυμόμενος άλλες δύσκολες διαπραγματεύσεις, ε, έχω συνηθίσει ένα τέτοιο κείμενο διαβάζω τουλάχιστον πέντε φορές πριν αποφευθώ. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος. Κατά βάση όμως παραμένει μια δομή σε κάποια στοιχεία. Έχει δίκιο η συνάδελφος Κρέσλε δεν θέλει κανένας να βρίσκεται στη θέση της ΥΠΑ της εκπροσώπου ή του νέου Γενικού Διευθυντή. Και οπωσδήποτε υπάρχει και κάποια ανακατοσούρα, μου επιτρέπει να το πω έτσι, στις ε, δομές που προτείνονται. Θα πρέπει λοιπόν η αναθεώρηση και ο έλεγχος να παίξουν ε, ρόλο. Αυτά που είπαν ο συνάδελφος Γκάιου και ο συνάδελφος Φάρμ είναι πραγματικά οι βασικές σκέψεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια στις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου διαφο... υπάρχει διαφορετικός τρόπος εργασίας. Υπάρχουν επιτροπές που δεν υπήρξε ακόμα ποτέ ε, Άλλε Άλλες όμως... Ε, επιτροπές όσον αφορά τις ε, εντολές και λοιπά έχουμε εργαστεί με μία ένταση που δυστυχώς δεν υπάρχει πάντα και ούτε σε νομοθετικές επιτροπές ε, του σώματος. Ίσως λοιπόν εμείς είμαστε πολύ επικριτικοί όσον αφορά την εργασία άλλων επιτροπών. Από την άλλη μεριά, αν κοιτάξουμε τις δυνατότητες ε, για να συμβάλλουμε σε αυτά, βλέπουμε ότι εμείς εδώ δεν έχουμε συναπόφαση, αλλά πρέπει να γνωμοδοτήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς λυπούμε ότι το ένα θέμα προωθήθηκε ταχύτατα και το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν προώθησαν τα άλλα στοιχεία της δέσμης έγκαιρα και εδώ ε, φαίνεται ότι θέλουν να μας φάνε, όπως σας είπα, μπουκιά, μπουκιά. Θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν και όσον αφορά την ε, διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των βουλευτών. Και θα πρέπει να σκεφτούμε Τι θα σημαίνουν όλα αυτά όσον αφορά την πρόθεση διαδικασίας, πράγμα που είναι δύσκολο. Εάν έχουμε κατόπιν διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό, εάν έχουμε κατόπιν διαπραγματεύσεις για το πώς θα οργανωθεί ένα τμήμα του δημοσιονομικού κανονισμού που ασχολείται με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ξέρουμε όλοι τι θα γίνει. Η πίεση θα συνεχίσει να αυξάνεται και εγώ δεν θέλω να αναλάβω ευθύνη όταν τελικά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο ορισμένες επιτροπές του Κοινοβουλίου εδώ σηκωθούν και πιέσουν να περάσει διορθωτικός ε, προϋπολογισμός υπό κάποια συγκεκριμένη μορφή και μετά θα πρέπει να αποφασίσουμε για την επαναχρήση των κονδυλίων. Με δύσκολο τρόπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για το τι θα γίνει στους επόμενους μήνες στο σώμα εδώ και κατά πόσο τελικά θα έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε. Γιατί θα πρέπει ίσως να πάρουμε κάποιες προκαταρτικές αποφάσεις γιατί για πολλές διαπραγματεύσεις δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρεύουμε όπως το θέλουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και δεν ξέρω αν θα πετύχουμε το στόχο μας με το να πάρουμε μια τέτοια απόφαση τον Ιούλιο ή όπως θέλουν πολλοί να αναβάλουμε και να περάσουμε σε μια κανονική διαδικασία. Γιατί ε, εάν το, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θέλουν, μπορούμε σε δύο εβδομάδες να τελειώσουμε. Αλλά δεν θέλουν, δεν μας δίνουν τίποτα. Το είπαμε και το ξαναείπαμε στο παρελθόν, το ζήσαμε σκληρά και άσχημα στο παρελθόν και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, το να συμφωνήσουμε αυτή τη στιγμή ε, στα γρήγορα μία δομή για την ε, υπηρεσία εξωτερική δράση και να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε γι' αυτό, αναξίζει λέω τον κόπο με το να περιμένουμε και να πάρουμε μία καλή και βασική, βάσιμη απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μπέκε. Έχει έρθει και ο κύριος Μπρουκ, Μπροκ βάλλον για να υποστηρίξει και να μας πει και κάποια παραπάνω από αυτά που ε, είπε ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Γκαρίγα Πογέδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ θεωρητικό. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, Μπέγκε. Το πρόβλημα δεν είναι σε αυτά που μας παρουσίασε ο κύριος ε, Γκουαλτιέρη. Ε, σαφώς θα υπάρξουν και σωστές τροπολογίες με τις ε, γλωσσικές μετατροπές που πρέπει. Θα έχουμε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο σαφώς θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει βέβαια είναι μια εις βάθος συζήτηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τις ευαισθησίες από τις διάφορες επιτροπές και αυτή η εις συζήτηση δεν έχει γίνει ακόμα. Εάν μπορέσουμε να την κάνουμε από τώρα μέχρι να κλείσουμε για τον Ιούλιο, καλό θα ήταν. Αλλά το βασικό για μας που είμαστε μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών εξακολουθούν να είναι το ερώτημα ποια είναι η επίπτωση στον προπολογισμό για αυτή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι ο διορθωτικός προπολογισμό παριθμών 6, ο οποίος παρουσιάστηκε χθε και για τον οποίο θα μιλήσουμε το Σεπτέμβριο, αλλά το ποια είναι η σχέση του προπολογισμού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ε, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα και τι επιπτώσεις θα έχει στις ε, παρούσες δημοσιονομικές προοπτικές. αν ο προπολογισμό ε, θα είναι συμβατός με το παρόν πλαίσιο, αν θα πρέπει να το εισεγάγουμε στην αναθεώρηση της ε, πολιετούς προσαρμογής που προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο. Δηλαδή, από πλευράς προπολογισμού θα πρέπει να περιμένουμε την πλήρη αξιολόγηση του προπολογισμού αυτής της εξωτερικής υπηρεσίας ε, ε, εξωτερικής δράσης για να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουμε στις ε, πολιετές δημοσιονομικές προοπτικές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί στην έκθεση Μπέγκε είναι πολύ δύσκολο οι πολιτικές ομάδες να παρουσιάσουν την άποψή τους χωρίς να γνωρίζουν πόσο ακριβώς θα μας στοιχήσει αυτή η εξωτερική υπηρεσία και τι επιπτώσεις θα έχει για τις υπόλοιπες ε, γραμμές προπολογισμού και τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Μέχρι να διασκεδαστεί αυτή η αμφιβολία μπορούμε να εγκρίνουμε μία σειρά από εκθέσεις, να λέμε ότι προασπίζουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, αλλά από πλευράς προπολογισμού θα είναι τα πάντα απολύτως απροσδιόριστα μέχρι να έχουμε απτά στοιχεία, ποσά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαρίγκα. Επειδή ήρθε ο κύριος Μπροκ, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ο κύριος Γουαλτιέρη μας παρουσίασε αυτά τα οποία διαπραγματευτήκατε και συμφωνήσατε χθες στη Μαδρίτη. Κάποιοι εδώ στην Επιτροπή Θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή του Κοινοβουλίου σε σχέση με το αρχικό κείμενο που μας παρουσίασε το Συμβούλιο. Κάποιοι άλλοι ανησυχούν ότι η απόφαση η οποία προτείνεται να ληφθεί τον Ιούλιο για την έκθεσή σας είναι βεβαιασμένη και το Κοινοβούλιο δεν είχε τη δυνατότητα να εξετάσει και τα τέσσερα έγγραφα που σχετίζονται με αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτές λίγο πολύ είναι οι απόψεις. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, να μας δώσετε κάποια επιπλέον πληροφορία για τα όσα διαμήθησαν εχθές. Ε, Ευχαριστώ. Επικίνδυνο άσκηση στο σκηνή είναι αυτή που κάνω, γιατί πρέπει να πω κάτι για πράγματα που δεν ξέρω, αλλά βέβαια συνήθως κανένας μπορεί πιο πολλά να πει για αυτό που δεν ξέρει παρά για αυτό που ξέρει. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Δεν θέλω να επαναλάβω την επιτυχία παρουσίαση που έκανε ο κ. Καλτιέρη ήδη. που βασίζεται στις γνώμες που έχει αυτή η Επιτροπή. Ενδυναμώνονται τα δικαιώματα της κοινότητας μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα σαν κοινοβούλιο την ε, ε, Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης και πολιτικά, όχι μόνο δημοσιονομικά. Και το θέμα, μια που οι λειτουργικοί προβλησμοί παραμένουν πάντα στα χέρια της ε, Κομισιόν, δεν αλλάζει τίποτα. Και νομίζω ότι εξασφαλίζεται το πιο σημαντικό που θέλαμε. Όλοι ξέρουμε, ο καθένα μα θα είχε γράψει διαφορετικό κείμενο. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε ένα συμβιβασμό μεταξύ 3,5 θεσμικών οργάνων. Και θα πρέπει να δούμε ότι η επιθυμία που υπήρχε όλα να γίνονται σου στην Κομισιόν ήταν κάτι που δεν ακολουθούσε κανένας, ε, κανένα κράτος μέλος και έτσι θα πρέπει να επανέλθουν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου διαφορετικά και αν δεν το καταφέραμε ή δεν το καταφέρουμε δεν θα έχουμε καμία υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και το θέμα είναι ότι αυτό με τα δύο καπέλα και την εξωτερική υπηρεσία εξωτερική δράση είναι δική μας ιδέα για να μπορέσει έτσι να παίξει σημαντικό ρόλο μέσα στη διεθνή κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε τελικά να αποδείξουμε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που οδηγούν οι σημεία των αρμοδιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία δεσμευτική απόφαση πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Πολλοί το μελέτησαν και που εξετάζουν την κατάσταση στο Συμβούλιο και οι οποίοι λένε ότι εάν ξανανοίξει η δέσμη και υπάρχουν καθυστερήσεις, τότε ορισμένες χώρες θα συμπεριθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε χειρότερη κατάσταση από ό,τι πριν. Ή θα έχουμε μια υπηρεσία τύπου υπηρεσία Σολάνα, που δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς. Και θα πρέπει να δούμε ότι στο τομέα διαβούλευσης δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να προφυλάβουμε μέχρι τη σύνοδο του Ιουλίου. Άκουσα τι είπε και ο κ. Γκαρίκα. Αυτά είναι δυνατά μόνο εάν βάσει συζητήσεων στις πολιτικές ομάδες οι πολιτικές ομάδες ε, το δώσουν να δείξουν ότι είναι δυνατό. Ωραίο θα ήταν να τα καταφέρουμε τον Ιούλιο. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια ευρεία πλειοψηφία που είναι πιο σημαντική από το αν βιαστούμε. Θα πρέπει λοιπόν τις επόμενες 8 μέρες να κάνουμε μία αξιολόγηση. Σήμερα και αύριο έχουμε τη συζήτηση στις δύο επιζουσίες αρμόδιες επιτροπές και μετά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ήμουν μόλις τώρα στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Τα πράγματα έδειχναν καλά. Γιατί πολλά πετύχαμε για την ε, πολιτική ανάπτυξη στο τομέα αυτό. Υπάρχουν και εκεί επικρίσεις, θα έπρεπε κάτι να γίνει διαφορετικά, κάτι να έχει ενταχθεί κάπου αλλού. αλλά θα μπορούσαν να συμφωνήσουν και με τη δικασία για τον Ιούλιο. Αυτό βέβαια θα είναι απόφαση των πολιτικών ομάδων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία που να εξασφαλίζει επαρκή συζήτηση. Δεύτερον, απορρίψαμε ρητά να υποχρεωθεί το Κοινοβούλιο να εξτάσει το θέμα τον Ιούλιο. Απορρίψαμε ρητά να αναλάβουμε την υποχρέωση σχετικά με το τι θα κάνουν οι διάφορες επιτροπές με την έκθεση αυτή, δύο με την ε, έκθεση συναπόφαση. Αυτό είναι μια τελείως ανοιχτή διαδικασία, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση και είμαι σίγουρος ότι όσον αφορά τη διαδικασία συναπόφασης για το κανονισμό του προσωπικού δεν θα αποφασίσουμε τον Ιούλιο. Και αυτό δεν είναι προϋπόθεση για την πραγματική θέση ισχύ. Το ίδιο ισχύει και για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Αν δεν υπάρχει τροποποίηση του άρθρου 1, όλα αυτά λένε περιτά. Μια λέξη να λείπει, τελείωσε. Γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα εκτός της Κομισιόν, σε περίπτωση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι με διαδικασία συναπόφασης δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία τον Ιούλιο, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα θέματα που θεωρούμε ότι σχετίζονται με τον συμπληρωματικό προεκλογισμό του 2010 σχετίζονται πολύ λίγο με την πολιτική συμφωνία πλαίσιο. Και όσον αφορά τις αποφάσεις αυτής εδώ της Επιτροπής για τον προπολογισμό δεν βλέπω να υπάρχει πίεση. Θα πρέπει να κάνει κανένα ό,τι θέλει. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και έχουμε καλούς λόγους το θέμα αυτό να το προσθέσουν και εάν δεν είναι ουδέτερο όσον αφορά τον ε, προπολογισμό, ε, αυτό που θα ενταχθεί είναι το κόστος των εθνικών υπαλλήλων. Και αν είναι το κόστος των εθνικών υπαλλήλων δεν πρέπει να υπολογιστεί αυτό κάπου στα ε, κονδύλια του Κοινοβουλίου. Μια που εγώ πριν από 25 χρόνια εγκατέλειψα αυτή την επιτροπή εδώ, εσείς έχετε εντωμεταξύ βέβαια πολύ περισσότερες πρακτικές εμπειρίες στο τι θα πρέπει να κάνετε. Αλλά νομίζω ότι βάσει της δέσμης αυτής ε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα να προωθήσουμε τον ρόλο της Ένωσης στον κόσμο. Thank you very much, uh, Mr. Brock. Before giving the floor... Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπουαλτιέρη για να κλείσει τη συζήτηση, και να μας δώσει τις δικές του εντυπώσεις, να μου επιτρέψετε να κάνω δύο παρατηρήσεις. Δεν είναι πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα της εξωτερικής υπηρεσίας. Περιμέναμε όλες τις προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις πήραμε πρόσφατα και αποφασίσαμε ότι θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή, αυτή στιγμή είχαμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας. Κάτι το οποίο φαίνεται να συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, υπήρξε μια εντατική προσπάθεια στα πλαίσια του τετραμερούς διαλόγου και από ό,τι φαίνεται σχετικά με την πρώτη επιλογή έχουμε πετύχει αρκετά καλά αποτελέσματα, ίσως όχι στα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα θετικά στοιχεία. Έχουμε λοιπόν τέσσερα έγγραφα. Το πρώτο είναι η έκθεση πλαίσιο, Brock η υπεύθυνη επιτροπή είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και εμείς θα δώσουμε απλά μια γνωμοδότηση. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας δεν έχουμε δυνατότητες συναπόφασης. Έχουμε τρεις άλλες αποφάσεις στις οποίες έχουμε τη δυνατότητα συναπόφασης, τον υπαλληλικό κανονισμό και τον δημοσιονομικό κανονισμό για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων. Εδώ υπάρχουν αρκετές ανησυχίες και λογικές ανησυχίες και ακούστηκαν. Θα είμαστε άραγε σε θέση να υπερψηφίσουμε την πρώτη έστω έκθεση τον μήνα Ιούλιο, την έκθεση πλαίσιο. Εγώ σέβομαι αυτά τα οποία είπατε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να μειώσω κανέναν, μάλλον θα αποφασιστεί από τις πολιτικές ομάδες το αν δηλαδή θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο θέμα τον μήνα Ιούλιο. Αυτή τη στιγμή θα αποφασιστεί στις πολιτικές ομάδες, οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους και τις συνέπειες του αν δεν ψηφίσουμε ή του τι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε επιπλέον αυτών που έχουμε ήδη πετύχει γιατί αυτό είναι ουσιαστικά ο μοναδικός λόγος για την αναβολή της ψηφοφορία τον μήνα Ιούλιο. Εάν λοιπόν οι πολιτικές ομάδες αποφασίσουν ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, θα το λάβουμε υπόψη μας και η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων θα προετοιμάσει μια γνωμοδότηση και εμείς από εκεί και πέρα δεν έχουμε σαν Επιτροπή προπολογισμού. από το να θέσουμε μία προθεσμία πριν από την ημερομηνία συζήτηση στην ΑΦΕΤ, στις εξωτερικές σχέσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας προτείνω λοιπόν, είναι μιας και έχουμε το έγγραφο μπροστά μας, που μας προτείνει ο Ρομπέρτο, και μιας και περιμένουμε να ληφθεί η απόφαση για το τι θα γίνει τον Ιούλιο, εφόσον συμπεριληφθεί τον Ιούλιο να θέσουμε μία προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και να χρειαστεί να υπάρξει και μία έκτακτη συνάντηση α, της Επιτροπής μας η οποία θα αποφασιστεί όμως από τον Πρόεδρό μας, τον κύριο Λαμασούρ. Αν αποφασιστεί ότι θα αναβληθεί η ψηφοφορία μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο, τότε δεν υπάρχει κάποιος επίγον χαρακτήρας και μπορούμε να συνεχίσουμε με τις κανονικές εργασίες μας. Αυτά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις διαδικαστικές, για τις διαδικαστικές εξηγήσεις των συνάδελφων Καλφίν. Εγώ αυτό το οποίο προτείνω είναι όχι να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, αλλά να μην αποκλείσουμε την δυνατότητα να ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να πάρουμε μία απόφαση η οποία θα πρέπει να είναι πολιτική απόφαση σε υψηλότατο επίπεδο την οποία θα λάβουν οι μεγάλες πολιτικές ομάδες σίγουρα. Θα πρέπει όμως να κρατήσουμε ανοιχτή την δυνατότητα έτσι ώστε οι πολιτικές ομάδες να έχουν δύο επιλογές. Αυτό επιβάλλει να υπάρξουν ορισμένες τεχνικές ρυθμίσεις οι οποίες ε, δεν είναι χωρίς προηγούμενα. Μπορούμε λοιπόν να περιοριστούμε αν θέλετε στο να συντονίσουμε μια διαδικασία η οποία να επιτρέπει την υιοθέτηση της εκθέσεως Φερχόσταυ Μπρόκ τον Ιούλιο εάν αυτό αποφασιστεί εκεί όπου θα αποφασιστεί. Επί της ουσίας τώρα. Η κυρία Τρούπελ έφεσε ένα ερώτημα πάνω σε ένα θέμα στο οποίο σε επίπεδο πόρων εννοώ είμαστε αρμόδιοι και δεν ανήκει θα έλεγα σε, στη συνολική έκθεση στην οποία εμείς δεν έχουμε παρασυμβουλευτικό ρόλο. Στα πλαίσια λοιπόν της κανονικής, της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας υπάρχει η πρόταση του προϋπολογισμού που έχει γίνει Είναι κάτι το ξεχωριστό της συζήτησης που γίνεται ειδικά για την έκθεση Μπροκ. Θα αξιολογήσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση στα πλαίσια της τακτής δημοσιονομικής διαδικασίας. Για την παρατήρηση του κυρίου Μπέγκε. πάντα είναι χρήσιμο να έχει κανείς περισσότερο χρόνο και να κάνει περισσότερες συζητήσεις. Αλλά σχετικά με την πρόταση του δημοσιονομικού κανονισμού, έχει παρουσιαστεί εδώ και τρεις μήνες αν δεν κάνω λάθος, ο κανονισμός για το προσωπικό στις αρχές Ιουνίου έχει δημοσιευθεί, αν και είχαμε τα στοιχεία εδώ και αρκετούς μήνες. Και να πω ότι οι όροι με τους οποίους συζητάμε την εξωτερική αυτή υπηρεσία είναι γνωστοί εδώ και αρκετό καιρό. Είναι ένα σημαντικό θέμα, έχει προεκτάσεις και δεν είναι απλά θα έλεγα κάτι το οποίο επαναλαμβάνει τη διαδικασία του Οκτωβρίου 2009 με την έκθεση πρωτοβουλίας. Έχει ξεκινήσει η κανονική λοιπόν κοινοβουλευτική διαδικασία για την έκθεση Μπρόκα, αλλά λόγω μία συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής. Του να λάβουμε δηλαδή υπόψη ότι πρόκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση για μια διαδικασία διαβούλευσης. Και ότι το θέμα είναι ο χρονισμός περισσότερο παρά το ίδιο το περιεχόμενο της έκθεσης. Θα μπορούσαμε βέβαια, μιας και συζητάμε αρκετό καιρό ε, την έκθεση Μπροκ, να την είχαμε ήδη εγκρίνει και η καθυστέρηση αυτή ίσως και να μας αποδυναμώνει τελικά. Πάντως η δυνατότητα που έχουμε μπροστά μας ανάμεσα στις διάφορες άλλες διαδικασίες που είναι διαθέσιμες, ισχυρές πολιτικά, η πρόταση αυτή είναι η πιο καλή, δηλαδή πια μία πρόταση η οποία τώρα βασίζεται στη συμβιβαστική λύση η οποία από ό,τι φαίνεται για το Συμβούλιο είναι πιο προχωρημένη από όσο θα επιθυμούσε, αλλά δεν αμφισβητεί αν θέλετε τις κανονικές διαδικασίες, τις νομοθετικές και τις δημοσιονομικές διαδικασίες, οι οποίες καλύπτουν τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σωστή διαδικασία. Μπορεί κανείς να επιλέξει και διαφορετικές ατραπούς, αλλά εν πάση περιπτώσει σχετικά με το επιχείρημα του κυρίου Μπέργκε υπάρχει και ο αντίθετος κίνδυνος. Ουσιαστικά δηλαδή να απορριφθεί η συμβιβαστική πρόταση και να φτάσουμε σε μία υιοθέτηση της έκθεσης Μπροκ το φθινόπωρο, μέσα σε ένα πολιτικό κλίμα σαφέστατα επιβαρημένο, αλλά και κάτω από μια πολύ ισχυρή πίεση έτσι ώστε να καταλήξουν όλες οι νομοθετικές διαδικασίες. Αυτό θα μας αποδυναμώσει. Και για τα υπόλοιπα θέματα και για τα άλλα και όχι μόνο για την έκθεση Μπροκ. Εν πάση περιπτώσει οι πολιτικές ομάδες με τον δικό τους δημοκρατικό τρόπο θα λάβουν τις αποφάσεις που πρέπει. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο σας ζητώ είναι να αφήσετε ανοιχτή την δυνατότητα να γίνει η έκθεση προκδεκτή τον Ιούλιο. Είναι μία από τις κανονικές δυνατότητες τις οποίες έχουμε για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουαλτιέρη. Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τη συζήτηση για σήμερα λήξασα. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή λοιπόν. Εάν αποφασιστεί να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, θα προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα μας αναλόγως ώστε να έχουμε την γνωμοδότηση νωρίτερα. Αυτό θα ανακοινωθεί στη συνέχεια στους υπολείπους. Επειδή έχουμε καλύψει όλα τα σημεία της ημερήσιας ε, διάταξης, να πω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 13 Ιουλίου, 13 και 14, αν δεν υπάρχει ε, κάτι επίγον το οποίο